Okay, good morning everybody. Um, Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα αρχίσουμε με το σημείο 16 που είναι πολύ σημαντικό που αφορά την έκθεση κοινωνικής προστασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, οπότε δυστυχώς ε, δεν έχω ακόμη διαβάσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι μοναδική στον κόσμο γιατί δίνει μια παγκόσμια θεώρηση της κοινωνικής προστασίας και της εκτιμήσεις ε, της ασφαλιστικής κάλυψης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολλές φορές συζητήσει πολύ για τη σημασία της οικουμενικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αν θέλουμε αξιοπρεπείς κοινωνίες πρέπει να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας ελάχιστο σε όλες τις χώρες και νομίζω ότι η προσκεκλημένη μας θα μας πει κατά πόσο αυτό είναι δυνατό και αν ε, προχωρούμε ή παναχωρούμε υπάρχει πάρα πολύ πίεση στους προϋπολογισμούς. Λόγω της κρίσης του 2008 εμείς είδαμε την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μου να υπαναχωρεί σε μεγάλο βαθμό. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και τι γίνεται στις χώρες εταίρους μας. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και λόγω των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, γιατί το καλοκαίρι το... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει προτάσεις για την... Ε, τον επόμενο γύρο δαπανών για τα επόμενα 7 έτη, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον Ιούνιο θα γίνει μια δημοσίευση των, προγραμμάτων, των νέων προγραμμάτων. Οπότε θα συζητήσουμε πώς πρέπει να είναι τα νέα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας με τους εταίρους μας ε, και η κοινωνική προστασία μπορεί να είναι κάτι που θα είναι σημαντικό στο πλαίσιο των νέων αυτών προγραμμάτων. Οπότε, Καλώς ήρθατε κυρία ορτή. Ε, με πολύ χαρά περιμένουμε να δούμε τι θα μας πείτε. Θα δείτε την παρουσίαση της ε, προσκεκλημένη μας στο Στι οθόνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να, είναι εδώ, να είμαι εδώ σήμερα, να σα παρουσιάσω αυτήν την έκθεση κοινωνική προστασίας. Είναι προϊόν ε, δουλειά ε, τριών χρόνων συλλογής δεδομένων από διάφορες χώρες. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ να σα δείξω τα αποτελέσματα αυτής τη έκθεση. Μου φαίνεται ότι δεν δουλεύει όμως το τηλεκοντρόλ μου και δεν μπορώ να αλλάξω τις ε, διαφάνειες. We'll just have a little while we resolve the technical problem. okay, I, I I continue because I understand it's very limited time. No, no, you're fine. Ε, με το χρόνο δεν έχετε πρόβλημα, εντάξει. Μισό λεπτό να μας, το, να μας βοηθήσει ο, ε, η συνάδελφος. Α, να σας δώσω το τηλεκοντρόλ. Πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα αν θα δουλέψει. Είναι αρκετά Ωραία. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη παρουσίαση. Ε, δεν θα διατρέξω όλες τις διαφάνειες, αλλά σας δίνει τα μηνύματα κλειδί για να κατανοήσετε την πολιτική και τα βασικά συμπεράσματα. Τώρα, ε, ε, έχουν εγκριθεί, έχουν εγκριθεί τα σχήματα αυτά από τις, τα Ηνωμένα Έθνη. Το SDG 1-3 είναι τμήμα της ε, δράσης ε, καταπολέμησης της ε, φτώχειας προκειμένου να εκπονηθούν εθνικά μοντέλα με Καταπολέμηση της αξίας και ε, της Συμπεριλαμβάνουν τα κατώτατα όρια κοινωνικής ε, προστασίας. Και το 2000, από το 2013 να παράσχουν συνδρομή στους ε, φτωχούς. Ο δείκτης είναι η κάλυψη της κοινωνικής ε, προστασίας ε, σε όλη τη διάρκεια ζωής, δηλαδή για τα παιδιά, για τη μητρότητα, για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Όλα, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί και βασίζεται στην, ε, στον δίκτυο για την κοινωνική προστασία. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο το οποίο υπάρχει από το 1949 και αποστέλλεται σε διάφορες χώρες οι οποίες ε, απαντούν ε, συλλέγεται ε, σε περιοδικά διαστήματα και έχει προσαρμοστεί στους στόχους της στρατηγικής ανάπτυξης και έχουν εγκριθεί από διάφορα αναπτυξιακά Ινστιτούτα. Η βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Κοινωνικής Προστασίας περιλαμβάνει αυτά τα δεδομένα. Και ε, μετράει τα, ποσοστά του, πλανητικού, ε, του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος ε, καλύπτεται από την κοινωνική προστασία. Είναι 45% του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο, στο βορρά και τον νότο, που έχουν ε, τουλάχιστον ε, ένα ευεργέτημα από την ε, κοινωνική προστασία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι 55% δεν έχουν απολύτως τίποτα. τώρα, το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, ξέρετε από το πώς το βλέπουμε. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος δείκτης, τον οποίο παρακολουθούμε για πολλά χρόνια και το στοιχείο κλειδί δεν είναι ότι γίνονται μόνο μεταφορές ε, ε, χρημάτων, αλλά υπάρχει κάλυψη από διάφορα μοντέλα, ε, νοσήλια, περίθαλψη κλπ. Αλλά από αυτά μόνο 29% του πληθυσμού καλύπτεται από αυτή την περιεκτική συνολική κοινωνική προστασία. 5,2 δισεκατομμύρια δεν καλύπτονται καθόλου από την κοινωνική ασφάλιση, αυτή τη συνολική κοινωνική ασφάλιση. Τώρα, 45% λοιπόν του πληθυσμού καλύπτεται από τουλάχιστον ένα, έχει μία κάλυψη, ένα ευεργέτημα της κοινωνικής προστασίας ε, στην ε, Αμερική, τη Βόρεια και την ε, Νότια καλύπτεται τουλάχιστον το, το, καλύπτεται 70% από τουλάχιστον ένα ευεργέτημα η υποσαχάρια Αφρική είναι περίπου 20% και συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια περιοχή που είναι η Μέση Ανατολή η οποία, από την οποία δεν έχουμε ούτε ε, τα μισά αξιόπιστα στοιχεία. Άρα λοιπόν απομένει πολλή δουλειά να γίνει. Τώρα, ο στόχος μας είναι να δούμε πώς ε, ε, κατανέμεται η κοινωνική προστασία και πού είναι τα ελλείμματα. Ορισμένοι λένε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένες χώρες έχουν κάνει τεράστιες πρόοδους ε, την τελευταία δεκαετία που υπήρξε μια έκρηξη σχημάτων κοινωνικής προστασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και όλες είναι αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν πετύχει μια καθολική κοινωνική προστασία. Και πραγματικά αυτό το γράφημα είναι ε, πολύ εντυπωσιακό γιατί δείχνει την έκρηξη που έχει συμβεί στην Κίνα. Στην Κίνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι σχεδόν ε, καθολική η κοινωνική κάλυψη. Αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικά θεαματικό και μοναδικό στην ιστορία. Ε, δηλαδή μέσω των ε, συνταξιοδοτικών σχημάτων ε, και των σχημάτων των μοντέλων κοινωνικής ασφάλισης έχουν σχεδόν καθολική κάλυψη. Αλλά υπάρχουν άλλες ε, χώρες, ακόμα και αφικρινικέ χώρες, όπου είχαν μια εντυπωσιακή ε, ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας. Κατά το ίμιση δηλαδή, καλύπτουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένε τέτοιε χώρε Τώρα, το πώς ε, είναι διαρθωμένη η έκθεση. Μας εξηγεί το πώς η κάλυψη τη κοινωνική προστασίας λειτουργεί για τις διάφορες περιοχές, του τις διάφορες περιοχές και τους διάφορους τομείς μάλλον, τις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Καταρχήν, ε, τα παιδιά, ε, άτομα με αναπηρίες, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι κλπ. Δεν πρόκειται να επισέλθω στα λεπτομερή στοιχεία εδώ. Μπορείτε να τα στο γραπτό κείμενο, αλλά θα ήθελα να σε εξηγήσω το σκεπτικό. πώς λειτουργεί το μοντέλο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρώτο τμήμα το οποίο περιγράφει την κάλυψη, δηλαδή πόσα παιδιά καλύπτονται στην ε, περίπτωση αυτή και βλέπουμε ότι είναι 35% ε, των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο από ε, κάποιο μέτρο κοινωνικής προστασίας και 35% λοιπόν των παιδιών καλύπτονται από κάποιο μέτρο.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 κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά σημαίνει ότι 65% δεν καλύπτονται καθόλου. Και έπειτα η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση σε σχέση με το πώ οργανώνονται διάφορα συστήματα κοινωνική κάλυψη ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί δεν κατανοούν ε, την έννοια τη κοινωνική προστασία. Δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ εργαζόμουν στη UNICEF για πολλά χρόνια και τα γραφεία τη UNICEF κάνουν πολλέ μεταφορέ χρημάτων για τα παιδιά συνειδητοποιούμε ότι η πλειονότητα των ε, μεταφορών χρημάτων πλαισιώνονται σε συστήματα κοινωνικής προστασίας. Ε, δεν είναι, γίνονται ε, τυχαία, αλλά πλαισιώνονται από ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να εντάξει ανταποδοτικά συστήματα σε μη ανταποδοτικά. Αυτή λοιπόν είναι η πλειονότητα των συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι οργανωμένα με αυτόν τον τρόπο. Και ε, στη συνέχεια έχουμε μία περιγραφή του κόστους, δηλαδή πόσο στοιχίζει για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα... Ε, αυτό το οποίο εμείς ε, είδαμε είναι... ότι ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού είναι παιδιά και στην πραγματικότητα μόνο 1,1% του ΑΕΠ ε, δίδεται για κοινωνική προστασία των παιδιών. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει πολύ σημαντική υποεπένδυση για τα παιδιά που θα πρέπει να αντισταθμιστεί με κάποιο τρόπο. And then you have Um, και μετά έχουμε ένα τμήμα του κειμένου που περιγράφει τις βασικές τάσεις. Ένα είδος παράλληλων παραλληλισμού στις τάσεις. Δηλαδή υπάρχει τεράστια ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή υπάρχει μια μαζική έκρηξη της κοινωνικής προστασίας καθώς και τα διάφορα κοινωνικά ευεργετήματα ε, και άλλες χώρες όπου υπάρχουν προσαρμογές ε, των μοντέλων αυτών λόγω λιτότητας, μέτρων λιτότητας και ε, εξυγένσης του προπολογισμού. Ε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό στο πλαίσιο της συζήτησης είναι να δούμε ότι μέτρα βαχυπρόθεσμης προσαρμογής δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ε, πρόοδο. Γιατί τελικά αυτά τα μέτρα προσαρμογής, δημοσιονομικής προσαρμογής, δείχνουν ότι είναι εντάξει λογισμό αλλά όσον αφορά την ανάπτυξη των ε, συστημάτων κοινωνικής προστασίας, εδώ υπάρχουν ε, ελλείμματα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε η βραχυπρότα, στοιχεία, η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη να μην έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε ε, εργαζόμενους, άτομα σε, στην ε, ηλικία εργασίας, η μητρότητα 43%, 41% γυναικών που έχουν παιδιά έχουν κάποια μορφή κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο ακριβώς της μητρότητας. Επίσης έχουμε προστασία ανέργων, η οποία είναι χαμηλή, 8% δεν καλύπτονται επίσης άτομα με αναπηρίες μόνο 28% ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες καλύπτονται από κάποια μορφή από κάποια μορφή ε, κοινωνικής προστασίας. Εδώ βλέπουμε ε, πώς είναι τα συστήματα. Οι τάσεις ε, παρομοιάζουν από τη μία χώρα στην άλλη, η Χιλή, Ουρουάη, έχουν για παράδειγμα συνολική κάλυψη για άτομα βαριές αναπηρίες, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που, λόγω των τάσεων λιτότητας έχουν σοβαρά ελλείμματα, τουλάχιστον πρόθεσμα Επίσης έχουμε ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας που αφορά τις συντάξεις και είναι το πιο και αν δούμε τη στάση 68% όλων των ανδρών και γυναικών του κόσμου παίρνουν κάποιο είδος σύνταξης. Δηλαδή είναι το πιο εξελιγμένο εργαλείο κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, το συνταξιοδοτικό. Ε, και βλέπουμε όσον αφορά την κατανομή, ε, ε, η καθολική κάλυψη είναι στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία, στην Αμερική 68% στη, στην Ασία Ελληνικό 55% και στην Αφρική περίπου 30% του πληθυσμού καλύπτονται από κάποια μορφή κοινωνική προστασίας και πάλι στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν καθόλου αξιόπιστα στοιχεία. Άρα λοιπόν είναι ο πιο εξελιγμένος τομέας αλλά υπάρχει ένα χάσμα στο εξωτερικό μεταξύ των δύο φύλων και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτό αφορά το ανταποδοτικό σύστημα, γιατί οι άνθρωποι, οι, άνθρωποι, άντρες, συγγνώμη, ε, εισφέρουν περισσότερο στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι εισφορές των γυναικών ε, δεν είναι συνεχείς. Τώρα, ε, οι δαπάνες για την ασφάλιση ανάλογα με το ΑΕΠ, τώρα όσο φέρεται, όσον αφορά τις χώρες που έχουν καθολικές συντάξεις ε, δηλαδή συντάξει για όλους ε, είναι ορισμένες χώρες τις έχουν αλλά οι περισσότερες χώρες έχουν ένα μεικτό σχήμα ανταποδοτικών μοντέλων ε, μαζί με κοινωνική συνδρομή για εκείνους που δεν παίρνουν καθόλου συντάξεις η Βολιβία, το Κυριαζιστάν, ε, Μαυρίκιο, η Μογγολία κλπ. Ε, και στην έκθεση δίδονται εξηγήσει για το ε, πώς διαμορφώνεται η πολιτική οικονομία σε αυτές τις χώρες και πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όταν τα αναλύει κανείς. Επίσης έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση που αφορά την αντιστροφή ε, σε σχέση με τις ε, ιδιωτικέ ε, συντάξεις. Στο παρελθόν υπήρξε από την Παγκόσμια Τράπεζα μια τάση ιδιωτικοποίηση των συντάξεων. Αλλά αυτή η ιδιωτικοποίηση των συντάξεων δεν δούλεψε στην πράξη. Τελευταία δεκαετία εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα και ασκήθηκε ανοιχτά κριτική στα ιδιωτικοποίηση των συντάξεων και έτσι λοιπόν πολλές χώρες ε, πάλι γίνονται τα συστήματα συντάξεων και πάλι δημόσια. Ε, η Αργεντινή, η Βολιβία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, η Πολωνία και πολλές άλλες χώρες ε, στρέφονται προς τα εκεί. Τώρα έχουμε άλλα κομμάτια που αφορούν την προστασία της υγείας και εδώ θα θέλαμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ, αστικής, μεταξύ υγείας στις αστικές και στις περιοχές της υπαίθρου. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι 56% του παγκόσμιου πληθυσμού της υπαίθρου δεν καλύπτεται από καμιά μορφή ε, περίθαλψης. Και βεβαίως αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί κατεπηγόντως. Η έκθεση τονίζει την σημασία της μακροπρόθεσμης περίθαλψης ε, ανάλογα και με τη γύρανση του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή μόνο 6% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει συστηματική πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη ε, περίθαλψη. Και όλες αυτές οι επενδύσεις στην υγεία και σε άλλους τομείς θα είναι τεράστια πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι ο τρόπος να το μιλήσουμε θετικά γιατί υπάρχουν, ε, γίνονται πολλές συζητήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση σαν ένα κόστος. Στην πραγματικότητα ε, πρόκειται για μια επένδυση γιατί δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Και αυτή τη στιγμή και υπάρχει ένα δυναμικό να προσλαμβάνονται ε, κοινωνικοί λειτουργοί ε, που θα ε, φροντίζουν ε, πολλές ομάδες του πληθυσμού. Τα παιδιά, για παράδειγμα. Ε, αυτή η διαφάνεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι ένας χάρτης του κόσμου και το πώς η κοινωνική προστασία αναπτύσθηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Ο πρώτος χάρτης που είναι σχεδόν λευκός εξ ολοκλήρου είναι γύρω στην αλλαγή του αιώνα, το 1900 και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μόνο λίγες ευρωπαϊκές πρωτοπόρες χώρες οι οποίες αναπτύσσουν κοινωνική ασφάλιση αλλά την εποχή εκείνη είχαν κάποια κοινωνικά ευεργετήματα κλπ. Και όσο περνάνε δεκαετίες διαπιστώνομαι ότι χρωματίζονται περισσότερο οι χάρτες. Πρόκειται λοιπόν για μια μακρά διαδικασία και το καθήκον όλων μας είναι πράγματι το 2030 να χρωματιστεί με πολύ έντονα χρώματα όλος ο χάρτης για να εξασφαλίσουμε ότι οι τάσεις αυτές που ε, εξελίχθηκαν με το πέρασμα των δεκαετιών οφείλεται ακριβώς το, στην μάχη που έδωσαν οι γονείς μας προκειμένου να κατοχυρωθούν συστήματα κοινωνικής περίθαλψης και αυτή, αυτός ο αγώνας θα πρέπει να συνεχίσει και σήμερα και αυτό είναι χρέος μας προς τις μελλοντικές ε, γενναίες. Μπορεί να κάνουμε προσαρμογέ για μικρό χρονικό διάστημα, πρόθεσμα αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μα την ευρύτερη εικόνα. Την ευρύτερη εικόνα ότι η κοινωνική προστασία για του πολίτε πρέπει να συνεχίσει γιατί εμείς είμαστε οι ΔΟΕ, έχουμε ένα τμήμα που αφορά την κύρωση των συμβάσεων που είναι σημαντικό για να μπορέσουν οι χώρες να ε, συνεχίσουν από μόνες τους και μετά έχουμε και την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι ε, από κοινού ε, είναι πώς θα καλύψουμε τα κενά. Να θυμόμαστε το 45% του πληθυσμού που καλύπτεται από τουλάχιστον ένα επίδομα και έχουμε 55% που δεν καλύπτονται από απολύτως τίποτα. Είναι λοιπόν απολύτω σαφέ ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην κοινωνική προστασία και αυτό είναι ένα ζήτημα πόρων, ένα ε, ζήτημα ε, βοήθειας και ένα ζήτημα εθνικών πόρων. Θα δούμε πιο μετά ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο ε, σε αρκετές χώρες Υπάρχει επίσης και το ζήτημα του προγραμματισμού των προγραμμάτων, του σχεδιασμού των προγραμμάτων. Έχουμε ε, ένα τμήμα του πληθυσμού που καλύπτεται από, ε, τους, ε, από την κοινωνική ασφάλιση και υπάρχει και ένα δίκτυο ασφαλείας κάτω-κάτω για τους στοχούς, αλλά το ενδιάμεσο κομμάτι λείπει εντελώς. Στην Αφρική, για παράδειγμα, όπου η κοινωνική ασφάλιση είναι λιγότερο ανεπτυγμένη, υπάρχει, ας πούμε, η κορυφή της πυραμίδας, άνθρωποι που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείε και που καλύπτονται από κοινωνική προστασία, άνθρωποι πάρα πολύ φτωχού με δίκτυα ασφαλείας και δεν δεν, αυτό που απουσιάζει εντελώς είναι ε, το ενδιάμεσο, το μεσαίο κομμάτι της ε, πυραμίδας. Εκεί είναι που πρέπει να ενισχύσουμε τις μεσαίες τάξεις, γιατί εκεί ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτοί που ανοίγουν επιχειρήσεις, είναι αυτοί που καταναλώνουν προϊόντα, είναι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν μια χώρα να λειτουργήσει. Αυτή η, το, αυτό το μεσαίο κομμάτι λοιπόν της πυραμίδας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνουν λοιπόν όλο και περισσότερο οι οργανισμοί είναι να προσπαθούν να νομιμοποιήσουν αυτοί που δουλεύουν στον άτυπο τομέα, δηλαδή σε ασταθείς δουλειές, χωρίς συμβάσεις εργασίας κλπ. Προσπαθούμε να, ε, προσπαθούν λοιπόν να νομιμοποιήσουν αυτές τις ε, ε, θέσεις εργασίας. Ζήσουν, ένα παράδειγμα στην Ουρουάη. Η Λατινική Αμερική είναι πρωτοστάτης και καινοτόμος σε πολλούς τομείς κοινωνικής προστασίας. Προσπαθεί δηλαδή ε, να έχει έναν φορολογικό συντελεστή στον οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή επιδότηση. Ένα, δύο, τρεις εργαζόμενοι που δουλεύουν άτυπα πληρώνουν έναν πάρα πολύ συμβολικό φόρο που είναι πάρα πολύ μικρός ε, και η κυβέρνηση επιδοτεί την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους συγκεκριμένους εργαζομένους και έτσι υπάρχει ένα τεράστιο αριθμός εταιριών που ε, επισημοποιούνται κατά κάποιο τρόπο ε, υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια στην έκθεση, αλλά αυτό είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα και ήθελα να το επισημάνω. Πρέπει να προσέξουμε ε, το εξής. Οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να υποφελούνται από αυτό το οικουμενικό σύστημα, οι άνθρωποι με AIDS, οι μετανάστες, ε, ε, πρέπει να δημιουργούμε κοινωνικά συστήματα προστασίας ε, σε ευάλωτα πλαίσια κλπ. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υποεπένδυσης στην κοινωνική προστασία, που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπετε τι, από γεωγραφικής απόψεως, τι επενδύουν οι χώρες στην κοινωνική προστασία. Βλέπετε το Βορρά, ο οποίος έχει πολύ περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και στον Νότο πολύ περιορισμένη επένδυση. Εδώ λοιπόν η αναπτυξιακή βοήθεια ειδικότερα στις χώρες οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, μπορούμε εμείς να παίξουμε ένα ρόλο. Τι κάνουμε ιδανικά. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα ε, και στη συνέχεια προσπαθούμε να σημειώνεται πρόοδο σε διάφορους τομείς. Ε, υπάρχουν οι δυνατότητες ε, επέκτασης ε, της δημοσιονομικής, της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ περιορισμένος ο προπολογισμός, δεν γίνεται σωστά η συλλογή των φόρων κλπ. Η Βολιβία, για παράδειγμα, πληρώνει ένα γενικό ε, επίδομα για τα παιδιά βάσει μιας πάρα πολύ μικρής φορολογίας ε, για την εξόριξη μεταλλευμάτων. Ε, μπορεί να γίνει δηλαδή φορολόγηση του εισοδήματος με διάφορους τρόπους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πόρους αυξάνοντας τις κοινωνικές εισφορές. Πολύ ωραία παραδείγματα έχουμε στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη, στην Τινησία και υπάρχουν και άλλοι πόροι οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν τη δυνατότητα, την ικανότητα των χωρών να συλλέγουν εισφορέ για τις κοινωνικές επενδύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, βοηθούμε τις χώρες κατά αυτόν τον τρόπο γιατί διαφορετικά υπάρχουν ε, ε, κάποια μοτίβα μιας κατάστασης εντελώς ε, αδιέξοδης η οποία δεν ε, προχωρά ε, καθόλου. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε τα κενά, προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση του εθνικού διαλόγου και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς του ΟΗΕ. Τριμερός συμμετέχουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, το Υπουργείο Οικονομικών και βλέπετε λοιπόν πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα και πού υπάρχουν και να. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία και με τι κυβερνήσει για να δούμε τι χρηματοδοτικές δυνατότητες υπάρχουν για την ενίσχυση αυτής της ε, κάλυψης, ε, τι ανθρώπινοι, τι οικονομικοί πόροι χρειάζονται και επίσης να υπάρξει και μια συμφωνία μια, επί μιας εθνικής στρατηγικής που θα οδηγήσει στη βελτίωση της κάλυψης και της χρηματοδότησης. Ο ΙΔΟ λοιπόν έχει λειτουργήσει σε 136 χώρες κατά τα τελευταία έτη. Έχουμε κάποιες, ε, ένα πρόγραμμα ορόσημο το οποίο καλύπτει έναν συγκεκριμένο αριθμό χωρών και περιοχών δεν είναι όμως ε, ζήτημα μόνο μίας ε, οργάνωσης. Όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε 12 χρόνια ακόμη στη διάθεσή μας για να αποτελέσει πραγματικότητα η κοινωνική προστασία για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ε, σύμφωνα με το θεματολόγιο ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ πού μπορείτε να έρθετε, σε πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιζαμπέλ, που μας έδωσες μία τόσο περιεκτική και πλήρη προσέγγιση, ε, συγγνώμη, θεώρηση της ε, κατάστασης. Ε, βλέπω ότι οι συνάδελφοι ήδη ε, θέλουν να πάρουν το λόγο. Μπορούμε να διανύμουμε την έκθεση αυτή στα μέλη. Έχουμε ένα αντίγραφό τη, ώστε να έχουν όλοι τι λεπτομέρειε της ε, παρουσίασης που μας κάνετε, της παρουσίαση που μα κάνετε. Δεν μπορούσα να δω όλα τα αριθμητικά στοιχεία λεπτομερώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να τα δούμε. Ο Νόμπετ Νόιζερ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ότιτς για την έκθεσή σας. Ähm, das war natürlich ähm, Βεβαίως ήταν ε, μια πολύ γενική επισκόπηση για τις ε, κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά στάνταρτς και την κοινωνική προστασία. Και θα ήθελα τώρα να τονίσω περισσότερο το δικό μας ρόλο στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Γιατί η έκθεση λέει ότι τα μεγαλύτερα ελλείμματα βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική. Εκεί ε, αναφέρατε κάποια πολύ θετικά παραδείγματα από χώρες όπως είναι η Μποτσουάνα ή το Κάπο Βέρδε ή η Τανζανία. Και εμένα θα με ενδιέφερε να μας πείτε σε ποιο βαθμό η έκθεσή σας επηρεάζει την αναπτυξιακή πολιτική από την πλευρά των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συγκεντρωνόμαστε όσον αφορά την αναπτυξιακή εργασία ε, επικεντρωνόμαστε σε υποδομές, σε εκπαιδευτικά συστήματα, συστήματα υγείας ε, για παράδειγμα και πιστεύω ότι τα συστήματα υγείας ε, έχουν πάρει προς. το ερώτημά μου είναι λοιπόν πώς προσπαθείτε σε σχέση με την έκθεσή σας να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να συμπεριληφθούν τέτοια θέματα στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διευρυνθούν τα κοινωνικά συστήματα στις λιγότερο ανεπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι το εξής, το πώς οι ενδιαφερόμενες χώρες αντιμετωπίζουν την έκθεσή σας. Ε, πιστεύω ότι αν μια χώρα παρουσιάζεται από θετικό πρίσμα, θα, θα είναι καλόδεχτη η έκθεση αυτή, αλλά πώς αντιμετωπίζετε χώρες που δεν υπάρχουν καθόλου πρόοδοι στην ανάπτυξη. Έχετε περισσότερες δυνατότητες να ασκήσετε επιρροή. Ε, εκτός από το να τις κάνετε να ντραπούν. Shame and blame. Ε, οι χώρες ε, που κατεπηγόντως χρειάζεται να πάρουν κάποια κοινωνικά μέτρα. Τι κάνετε εσείς με αυτές τις χώρες. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Νόρμπερτ. Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ γιατί μας δώσατε μια πολύ πλήρη εικόνα της κατάστασης για την κοινωνική πρόνοια σε όλο τον κόσμο και μεταξύ άλλων με εντυπωσίασαν αυτοί οι χάρτες που μας δείξατε ε, από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα. Το 1926 φτιάξαμε το σπίτι μας στο Ελσί και υπήρχε ένα κουτί ασφαλείας Ξέρετε γιατί. Το λέγανε πώ την box γιατί το 1926 δεν υπήρχαν συντάξει και άρα θα έπρεπε εκεί σαν κουμπαρά να αποταμιεύουν. Γι' αυτό λέγανε safe box, σαν χρηματοκιβώτιο. Και στο χρηματοκιβώτιο τελικά έβαλα ένα μπουκάλι whisky και το κάλυψα το χρηματοκιβώτιο με έναν πίνακα ζωγραφική. Ακόμα εκεί είναι. Πάντω άκουσα αυτές αυτές τις στατικές ιδέες δηλαδή πως περισσότεροι από την άτυπη οικονομία θα μπουν στην mainstream οικονομία, από την γεωργική, στην ε, ε, τρέχουσα οικονομία, την επίσημη, οπότε θα υπάρχει κοινωνική προνοία. Για πέστε μας τώρα, πού βλέπετε ε, τα μεγαλύτερα κενά, ποιος είναι ο πιο ουραγός, γιατί θα πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι η κοινωνική πρόνοια είναι το μέλλον της χώρας. Πώς, πώς μπορούμε να κάνουμε εκστρατεία για αυτή την ιδέα. Ίσως και εγώ θα μπορώ να υποβάλω κάποιες λέει η Πρόεδρος κατόπιν των όσων είπε και η Χέιντι. Α, για αυτό το τελευταίο που είπατε, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για τις χώρες μας, πολλές φορές βλέπουμε ότι τα αφεντικά, οι βιομήχανοι συνειδητοποιούν ότι αρρωσταίνουν οι εργάτες. Οι εργαζόμενοι. Ε, και τελικά έχουμε ε, το... Είχαμε τον τυφοειδή πυρετό, είχαμε πάρα πολλά θύματα και έτσι ξεκίνησε το, το σύστημα δημόσιας υγείας. Να λοιπόν πώς όλοι επηρεάζονται από όλα αυτά. Και θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, μας είπατε αυτό το ποσοστό της μη 55%. Μα α, φαντάζομαι ότι αυτό έχει ανωδική τάση. Γιατί στις πιο φτωχές χώρες έχουμε εκθετική αύξηση και μείωση του πληθυσμού στις πλουσιότερες. Επομένως, θα έχουμε αντίστοιχη διακύμανση αυτού του ποσοστού. Α, ιδίως στην Αφρικα που έχουμε αύξηση. Και βέβαια προσθέσει ενδιαφέρον ότι κάποιε χώρε όπω το Βέλγιο, η η Αγγλία έχουν καλύτερη κάλυψη από ότι οι πιο φτωχέ στην Αφρική. Αλλά τι γίνεται με χώρε που βρίσκονται σε συγκρίσιμο επίπεδο. Γιατί εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τη μια χώρα στην άλλη. αν και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Είπαμε για την Ουρουγουάη. Είπαμε η Λατινική Αμερική παρουσιάζει όπω φάνηκε και στις διαφάνειες κάποια πρόοδο. αλλά σε κάποιε άλλε τα πράγματα πάνε προ το χειρότερο. Γιατί πήγανε καλύτερα εκείνε τι χώρε στην αρχή λόγω τη ανόδου τη τιμή των εμπορευμάτων και τώρα πέσανε. Τι λέτε για τη Λατινική Αμερική. Επίσης, προβληματίζομαι και στρέφομαι στους συναδέλφους που ασχολούνται με την ΑΚΕ, όπω τον Όρμπερτ και τους άλλους. Μήπως θα μπορούσαμε αυτό να το συζητήσουμε στη συνέλευση ΑΚΕ με τους εταίρους. Κάνουμε κάποιες πρακτικές συζητήσεις και όχι θεωρητικές για τα ψηφίσματα κλπ. Να μας πούνε. Να μας πούνε για το θέμα αυτό. Γιατί για όλες τις φορές ισχύει αυτό. Πολλές φορές η τα κοινοβούλια και τα συνδικάτα έδωσαν όθηση στο να συγκροτηθούν και επιστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Να, πού πρέπει να στραφούμε και να αναδείξουμε το πώς και τι θα πρέπει να γίνει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 διάβασα κατόπιν και την έκθεση. Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι κάτι με εξέπληξε θετικά και από πολλές πλευρές. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη στον κόσμο όσο αφορά την κοινωνική πρόνοια. Είδα όμως ότι σε κάποιες σχετικά μεγάλες περιοχές και απλώς πληθυσμού και έκτασης έχουμε διάφορες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας που βαδίζουν καλά. Μας είπατε επίσης, μας είπες τέλος πάντων, ότι υπάρχουν δύο γραμμές πλεύσης διαφορετικές, τέλος πάντων αποκλίνουσες. Όμως, αυτό μπορούμε να το δούμε και παραδοσιακά ότι δηλαδή αποκλίνουν αυτές οι δύο πορείες, οι δύο γραμμές, αλλά για την άλλη μεριά ότι συγκλίνουν όσον αφορά τα αποτελέσματά τους. Γιατί πολλά, πολλά προχωράνε έτσι. Και πολλοί από εμά όμως από την άλλη μεριά σημειώνουμε γύρισμα Οπότε έχουμε αυτή την ε, ιδέα ότι η ισορροπία θα επέλθει με έναν αγώνα δρόμο προς τα κάτω, μα δεν είναι έτσι ίσως, γιατί ο πύχης ανεβαίνει. Οπότε έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμο προς τα κάτω, όμως ε, αυτό δεν, είναι στο, δεν πάει στο πηγάδι δίχως πάτο, γιατί ταυτόχρονα το επίπεδο ανεβαίνει. Οπότε όλη αυτή η προβληματική ότι όλα έχουν σχέση με το κοινωνικό ντάμπινγκ, όλο αυτό το επιχείρημα ε, ε, έρεται, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και αλλού στον κόσμο έχουμε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ε, δημιουργούνται συνταξιωτικά συστήματα, προστασία ανηλίκων υπάρχει, ε, παιδεία, σχολεία. Οπότε βλέπουμε ότι στον κόσμο μειώνεται η ανισότητα σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι πριν από λίγο. Ταυτόχρονα δε. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι οι ανεπτυγμένες χώρες, περισσότερες δηλαδή από τις δικές μας, τα σχετικά αντίστοιχα συστήματα θα πάνε χειρότερα για διάφορους λόγους, για λόγους κάποιων κρατικών πολιτικών, ας πούμε, οι πολιτικές ε, λιτότητας, οι διάφορες περικοπές, οπότε έχουμε επιδείνωση, αλλά και για άλλο λόγο. Γιατί η επασχόληση σήμερα δημιουργεί κάποιες δυναμικές που υποβαθμίζουν και χτυπάνε τα συστήματα πρόνοιας. Να, οι συντάξεις. και η Ισπανία. πως λένε και οι Εγγλέζοι, αυτή τη χώρα ξέρω. Αυτήν, για αυτήν συζητώ. Οπότε, βλέπουμε ότι η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη έκταση, γίνεται πιο συχνή. Οπότε και έχουμε συρρήγνωση του συνταξιδοτικού και των συντάξεων. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι Όσοι σήμερα είναι 30-40 ετών, αυτή η γενιά δηλαδή, ε, δουλεύουν, αλλά οι σφορές τους είναι ανάλογες του μισθού τους, που είναι πάρα πολύ χαμηλός. Η mini job στη Γερμανία κλπ. Επομένως, σε 15-20 χρόνια τα πράγματα θα έχουν έρθει ανάποδα. Για πέστε μας επομένως ο πλευράς ILO τι λέτε. Επίσης, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει περισσότερο στα αστιοεξωτικά παρά στα συστήματα υγείας. Έτσι κατάλαβα. Είναι και θέμα κατανομής του κόσμου σε αστικές περιοχές σχέση με την Ήπεθρο, οπότε η δεύτερη κατηγορία είναι ως επιτοπλίστων ε, ακάλυπτη. Πάει και η ισότητα, πάει και η οικονομική ανεξαρτησία επίσης. Επίσης, απ, το είπε η πρόεδρος, η Λίντα. Κάτι σας ρώτησε η Λίντα, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, γιατί κάποιε χώρε που βρίσκονται στην ίδια φάση και βαθμό ανάπτυξη έχουν κοινωνική πρόνοια σε μερικές περιπτώσεις ε, ξεχωριστή, αρκετά διαφορετική δηλαδή. θα πρέπει τώρα να σας πω ότι ιδεολογικά από την πολιτική μου ομάδα αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι είναι θέμα της κρατικής πολιτικής δεν, δεν, δεν είναι έολο το επιχείρημα, δεν υπάρχει εναλλακτική ότι όλα τα κυβερνάει η αγορά, ό,τι και να κάνουμε το είναι το ίδιο. Αυτό το επιχείρημα αποδεικνύεται έολο εκ των πραγμάτων. Και πάλι για την Ισπανία να σας πω ότι έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ας πούμε ίδιους σε διάφορες ιστορικές φάσεις αλλά κοινωνική πρόνοια ε, σφαιρική κάλυψη, καθολική κάλυψη υγείας, πολιτικές ισότητας, όλα αυτά, όλα αυτά σε διαφορετικές φάσεις ιστορικές με την ίδια ανάπτυξη απέδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Άρα θα πρέπει να δώσουμε αγώνα τόσο ώστε οι κρατικές πολιτικές να είναι τέτοιες ούτω ώστε ούτως ώστε σε ισοδύναμες, σε αντίστοιχες καταστάσεις οικονομικής ανάπτυξης να δίνουν διαφορετικές ευκαιρίες στον κόσμο. Πολλές ερωτήσεις υποβλήθηκαν, αλλά ο τελευταίος να είναι ο κύριος Γκέρντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω μια, ε, σύντομη, ένα σύντομο σχόλιο. Είμαστε πολυάριθμοι σε αυτό το κοινοβούλιο που προβληματιζόμαστε σε σχέση με την πρόσβαση στην κοινωνική ε, προστασία σε όλες τις χώρες. Καταρχάς είναι ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Το Μαλάουι καταφέρνει να δημιουργήσει ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας παρά το γεγονός ότι δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Ε, καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα αλληλεγγύης το οποίο έχει μία κάλυψη ανεπαρκή αλλά εν πάση περιπτώσει τη συμμερίζονται όλοι σε, αυτό το, σε αυτή τη χώρα. Στις ΗΠΑ δεν ήταν ζήτημα μέσων ε, η μη ε, κάλυψη, μη οικουμενική ε, κάλυψη. Ο Ομπάμα δημιούργησε ένα σύστημα που επέτρεψε σε περισσότερο κόσμο να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα σε πολύπλουσες χώρες που δεν είναι τέλεια και υπάρχουν συστήματα σε φτωχές χώρες που πάλι δεν είναι τέλεια. Αλλά υπάρχουν και στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες. Οπότε είναι ένα ζήτημα κοινωνικής, ε, συγγνώμη, πολιτικής βούλησης. Δεύτερος προβληματισμός ποια είναι τα εμπόδια που παρακολύουν την πρόσβαση στην ε, κοινωνική ε, ασφάλιση. Όταν μιλάτε για τους Κινέζους, για παράδειγμα, μας λένε ότι το να υπάρχει κοινωνική προστασία σημαίνει λιγότερη, μάλλον λιγότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο. Για ποιο λόγο δεν καταφέρνουμε να βρούμε περισσότερους πόρους ε, για τις ε, κοινωνικές δαπάνες και η απάντηση είναι ε, αν το κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση του επίπεδου ανταγωνιστικότητά μας. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα όπου θα υπάρχει εξουδετερώση ε, μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων στο G20 ε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στο G20 και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνει μια πρωτοβουλία για να τεθεί αυτό στην ημερήσια διάταξη. Στην κυρία Μέρκελ είχα στείλει μια επιστολή πριν από ένα χρόνο περίπου όταν ήταν πρόεδρος του G20 και τη ζητήσαμε να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη. Δύο μήνες έλαβα την απάντηση ότι ήταν πολύ αργά για να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι εκρηκτική. Η υπάρχει κατάρρευση στις κοινωνίες μας γιατί δεν μπορούμε να χειριστούμε αυτό το σύστημα, δεν καταφέρουμε να βρούμε λύσεις. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Ε, μου λέτε λοιπόν ότι δεν γίνεται αυτό. Εκείνοι που έχουν την ευθύνη πρέπει να οργανώσουν ε, ε, ένα, ε, μια, έναν, κοινωνικό διάλογο για να το πω έτσι. Ό,τι συζητούμε εμεί εδώ το συζητούν και στον Ταβό. Απλώ εκεί όσοι συμμετέχουν στη συζήτηση τα τελευταίε δεκαετίε έχουν κάνει τα πάντα για να μην φτάσουν σε αυτήν την, τη λύση που εγώ μόλι σα περιέγραψα. Χρειάζεται πολιτικό κουράγιο, χρειάζεται πολιτικό ε, ε, Δεν χρειάζεται να είμαστε αφελείς, αλλά μπορούμε να είμαστε... Να, να, να ε, ε, βρούμε τουλάχιστον τις λύσεις. Να δώσω στην κυρία Ορτής το λόγο να μας απαντήσει και μετά θα δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο για να απαντήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, όσο τις έχει στο μυαλό τις φρέσκες, καλύτερα να απαντήσει και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι ερωτήσεις, όλες, οπότε σας ευχαριστώ. Ελπίζω να απαντήσω εξίσου καλά. Με ρωτήσατε αν υπάρχει ζήτηση. Σε 136 χώρες ε, έχουμε αναλάβει δράση τα τελευταία χρόνια. Όλες οι χώρες μας ζητούν την παράταση των ε, προγραμμάτων αλλά και τη βελτίωση των ανταποδοτικών των συστημάτων. Συγγνώμη. Πολλές φορές υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότηση ζητήματα ανθρωπίνων πόρων, ε, προσωπικού. Ε, έχουμε λοιπόν μια ζήτηση που είναι δύσκολο να τη διαχειριστούμε. Κάποιο επίση με ρώτησε αν υπάρχει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γιούκεν Χούμερ είναι εδώ ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να τα απαντήσει καλύτερα από μένα, για την ώρα δεν έχουμε λάβει υποστήριξη από την Επιτροπή. Πολλές πολλές ερωτήσεις έχω λάβει. Φυσικά οι πολιτικές είναι σημαντικές και εμείς τονίζουμε τα καλά παραδείγματα, συνήθως έτσι ο ΙΕ λειτουργεί και δεν τονίζει του, τα κακά παραδείγματα, αλλά τα καλά παραδείγματα που μπορεί κανείς να τα ακολουθήσει. Και υπάρχουν πολλά από τη Λατινική Αμερική κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά υπάρχουν και πολλά από την Αφρική και την Ασία τώρα. Η τάση είναι η αύξηση της κάλυψης, όχι η μείωση της, ε, ανεξαρτήτως του πληθυσμού, γιατί υπάρχει μία έτσι έκρηξη συστημάτων ε, στις ε, ε, χώρες τις αναπτυσσόμενες. Αυτή είναι η τάση, η επέκταση των συστημάτων, η συνέχιση των συστημάτων, η επέκτασή τους και εμείς εκεί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πώς το κάνουμε αυτό. Όπως είπατε και πολλοί από εσά, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Γι' αυτό ακριβώς Συνήθως αρχίζουμε από τον, κοινωνικό, από τον εθνικό διάλογο, από τον εθνικό διάλογο που βασίζεται σε δεδομένα ώστε να μην γίνεται πολιτικοποίηση του ζητήματος. Μπορεί κανείς να δει ποια είναι τα βασικά κενά, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, να προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τους εργοδότες μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να συμμετέχουν. Τρία επιχειρήματα υπάρχουν σε γενικές γραμμές, τα αναφέρατε όλοι. Το θέμα της ε, ανάπτυξης ανάπτυξη και τη παραγωγικότητα, γιατί αν οι άνθρωποι είναι άρρωστοι ή ε, είναι πολλά μέλη τη οικογένειά του άρρωστα, δεν μπορούν να εργαστούν. Υπάρχει ένα ζήτημα ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης ε, προφανέστατα, γιατί όταν ο κόσμος τρέφεται καλύτερα ή μπορεί να πάει σχολείο, έχει και αυτό σημασία. Υπάρχει και ένα σημαντικό επιχείρημα που είναι πολιτικό και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Η μείωση της φτώχειας και της ε, ανισότητας σε πολλές χώρες ε, δεν είναι βιώσιμη και δημιουργεί πολλές πολιτικές εντάσεις. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στον πληθυσμό ένα βασικό επίπεδο κοινωνικής ε, ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι που το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Είχα πάει στην Τινησία πολύ πρόσφατα και εκεί η κυβέρνηση μου ζητούσε να τη βοηθήσω να, δημιου... να ε, αντιμετωπίσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί έκαναν πάρα πολλές περικοπές στην κοινωνική προστασία. Η Αραβική Άνοιξη έγινε ε, σε αυτή την χώρα προσφάτως και υπήρχε και αύξηση της τρομοκρατίας, την οποία τη βίωσε πολύ αυτή η χώρα. Πρέπει κάπως να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες είτε εξασφαλίζοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι δεν ε, ασχολούνται με πολιτική και ασχολούνται ε, μόνο με το οικονομικό κομμάτι και αυτοί οι άνθρωποι όμως, άνθρωποι είναι, ε, πρέπει να έρθουν και αυτοί στο τραπέζι του διαλόγου για να μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που άπτονται και άλλων πτυχών. Το να υπάρχει λοιπόν ένας ανοιχτό διάλογος, όλοι, όλες οι οργανώσεις Κοινωνία των πολιτών, ε, τα, του Υπουργείου Οικονομικών, οι εργοδότες, ε, είναι πολύ σημαντικό από τις περισσότερες χώρες τέτοιου είδους αιτήματα και κλήσεις λαμβάνουν. Θα ήθελα λοιπόν να με βοηθήσετε να το προχωρήσουμε αυτό. Και άλλα πολλά ερωτήματα μου θέσατε επί των λεπτομεριών. Διαφορά μεταξύ των χωρών υψηλών ε, εισοδημάτων και χαμηλών ε, είναι το επίπεδο επιδημάτων. Μιλάμε τώρα για την κάλυψη, για την ε, ασφαλιστική κάλυψη. Ε, υπάρχει όμως κόσμος με 50 λεπτά τη μέρα. Ε, με, με, με βοήθεια 50 λεπτά τη μέρα και άνθρωποι με σοβαρότερες συντάξεις. Υπάρχει και το θέμα λοιπόν του επίπεδου των επιδομάτων. Ένα ακόμη παρα, παράδειγμα, στην Αμήμπια για παράδειγμα, το 2015 το ίδιο πρόβλημα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάει λοιπόν εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι α, υπάρχουν αυτά τα δημοσιονομικά προβλήματα, εκεί όμως έχουν ε, ένα συνταξιοδοτικό σύστημα Οικουμενικό πίστευαν εκεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανέμεται η ανάπτυξη μεταξύ του πληθυσμού, οπότε θεωρείται ένα δικαίωμα η σύνταξη για όλους όσους γίνονται 65 ετών. Όλοι λοιπόν έχουν σύνταξη. Το 2015 όμως 35 ε, δολάρια το μήνα ήταν αυτή η σύνταξη. Ένα δολάριο το μήνα περίπου δηλαδή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μία από τις ε, συναντήσεις ε, αποφασίζει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια δημοσιονομικός προς, ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Ε, να μην κόψουμε τις συμβάσεις λοιπόν. Τεράστια ήταν η συζήτηση και τι έκανε η κυβέρνηση μετά από αυτή την τεράστια συζήτηση αύξησε την σύνταξη που είναι τώρα 72 δολάρια το μήνα. Βλέπετε ότι δουλεύει μερικές φορές η συζήτηση, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η δημόσια συζήτηση, αυτός ο διάλογος και είναι σημαντικό να είναι εκεί κανείς για να υποστηρίξει τις χώρες με αυτά τα επιχειρήματα τα οποία μόλις είπατε. Όχι να λέτε απλώς ότι οι κυβερνήσεις θα το κάνουν. Οι κυβερνήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν ανταγωνιζόμενα ζητήματα. Υγεία, μεταφορές, νερό, ε, άμυνα, ε, υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία ε, πρέπει να τα λύσουν. Ε, αυτά ανταγωνίζονται μεταξύ του. Εμεί ω αναπτυξιακοί εταίροι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, τονίζουμε τα κοινωνικά θέματα και την κοινωνική προστασία. Διαφορετικά πάνε κάτω-κάτω ε, στο κατάλογο των προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θεωρώ ότι το σε σχέση με το πρόγραμμα του IMF, ε, κάτι που συζητήσαμε και χθες, ε, που περιστέλλονται αυτές οι δαπάνες, Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να, να την παρακολουθήσει και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης γιατί υπάρχει μια συζήτηση εντός της Επιτροπής για τη συνοχή των διαφόρων ε, πολιτικών. Και σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, θεωρούμε ότι δεν είναι καλή, σωστή πολιτική το να δίνουν με το ένα χέρι και να παίρνουν τα χρήματα με το άλλο. Γιούργεν Χόμερ, εγώ ε, εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση ε, που αφορά το τμήμα μετανάστευσης και απασχόλησης. Ακούσαμε ότι η κοινωνική προστασία για την οποία εγώ είμαι επιφορτισμένος έχει, ε, έχει εξαφανιστεί από την ε, πονημία του τμήματος. Αυτό πληροφοριακά. Καταρχήν θα ήθελα να, πω, να ευχαριστήσω το ILO που προετοίμασε αυτή την έκθεση. Πραγματικά είναι μια τεράστια προσπάθεια αυτή που καταβάλατε τα τελευταία χρόνια. Ε, και είναι κάτι βεβαίως που αναμένουμε ε, οργανισμοί όπως ο δικός μας. Χρειαζόμαστε νέα επικυρωμένα δεδομένα για να μας παράσουν τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Τα βασικά στοιχεία τα οποία μας δείξατε επισημαίνουν το 55% του πληθυσμού που δεν καλύπτεται από κοινωνική ε, προστασία και το 17% και το ποστό εκείνων συγγνώμη, που, που είναι ανεπαρκώς ε, καλυμμένοι. Ε, Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν και κάποια λύματα στην έκθεση αυτή γιατί ε, και στον τρόπο λειτουργία του ΑΕΛΟ, αλλά και στα δεδομένα αυτά. Αυτά, γιατί πρόκειται για δεδομένα τα οποία τα έχουν ε, διαθέσει κυβερνήσεις. Ε, και ίσως θα έπρεπε να βελτιωθούν οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων. <coughs> Όσον αφορά το 70%, εάν το καταλάβαμε καλά, αυτή είναι μόνο μια νομική κάλυψη που σχετίζεται με τη Σύμβαση 102 και η οποία αναφέρει τα ευεργετήματα της κοινωνικής προστασίας. Αλλά δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί γενικά είναι εξαιρετικά, είναι ικανοποιητική για μας η έκθεση. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα που τέθηκε εδώ για το ρόλο της Επιτροπής, τι κάνει η Επιτροπή με την ε, ε, ψηλή ζήτηση. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο της κοινωνικής προστασίας. Η Ζαμπέλ είπε ότι οι συζητήσει υψηλού επίπεδου με το ΑΕΛΟ και την Επιτροπή ε, κατ' ουσία είναι ανύπαρκτα. Έχουμε μία σχέση συνεργασίας, αλλά η επίδραση της έκθεσης αυτής, της λήψης ε, αποφάσεων εκ μέρους της Κομισιόν ε, είναι λυπής. Για να απαντήσω αυτό το ερώτημα θα ήθελα να πω ότι έχουμε και μία άλλη έκθεση σε σχέση με την παγκόσμια αξιολόγηση της ε, υποστήριξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την κοινική προστασία μέσω εξωτερικής δράσης. Η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί από το δικό μας τμήμα, το έχουμε αποστείλει προς όλους και καλούμε εσάς και τους συνεργάτες σας σε, και σε άλλες παρουσιάσεις. Πραγματικά είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη μελέτη, γιατί η αξιολόγηση αυτή καλύπτει ε, ποικίλε χώρες και λέει ξεκάθαρα ότι οι επενδύσεις της Επιτροπής στην κοινωνική προστασία είναι κάτω από 1% του συνολικού προλογισμού, είναι εξαιρετικά ισχνή. Και ε, αυτό το ε, μήνα ε, είχαμε σημαντικά αποτελέσματα εκεί όπου υποστηρίξαμε κάποιες χώρες εταίρους με την, στο επίπεδο της κοινωνικής προστασίας. Βεβαίως αυτά όλα αφορούν περισσότερο την κοινωνική συνδρομή αν θέλετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιγότερο την κοινωνική προστασία έτσι όπως την εννοούμε εδώ στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να καλέσω εκείνους που ενδιαφέρονται να δουν τα θέματα αυτά. Γιατί οι προσεγγίσεις υποστήριξης μέσω του προπολογισμού είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί πρόκειται για έναν πολιτικό διαλόγου, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος και το ακούσαμε και εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Η πολιτική βούληση είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Υπό την έννοια αυτή προσπαθήσαμε αυτό το χρόνο και τον προηγούμενο ε, και θα το συνεχίσουμε και φέτος να προωθήσουμε από το δικό μας ε, τμήμα ένα σφαιρικό πρόγραμμα κοινωνικής, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα ε, κοινωνικής προστασίας το οποίο δεν θα είναι τμήμα του ετήσιου προγράμματος του προηγούμενου έτους θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας και να εξετάσουμε το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η κοινωνική προστασία στο επίπεδο της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, προκειμένου να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας. Ε, και κάτι άλλο. Βέβαια, η αναβάθμιση συνδέεται με κάποιο κόστος. Αλλά τα στοιχεία τα οποία πήραμε από μια μελέτη για την Αφρική ε, λένε 1,1% του ΑΕΠ ε, μπορεί να υποστηρίξει μια ένα ποσοστό κάλυψη 17%. Like, um... Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θέλατε να διορθώσετε κάποιες, ε, κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς. Η ομιλήτρια, ναι, είναι αλήθεια. Όλα αυτά βασίζεται σε μια μελέτη που απευθύνεται στις κυβερνήσεις. Είναι δεδομένα τα οποία αντλούνται από τις κυβερνήσεις, αλλά όχι αποκλειστικά από τη UNICEF επίσης, από την Παγκόσμια Τράπεζα και αυτά τα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται στην ε, μελέτη μας ή από οικονομικές επιτροπές στις διάφορες περιφέρειες, ε, τις αναπτυξιακές ε, τράπεζες κλπ. κλπ. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί για Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να προωθήσουμε την συνοχή των πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστούμε την Ιζαμπέλ Ορτής. Μας δώσατε μια πολύ ε, συμπεριληπτική ε, προσέγγιση, ε, περιεκτική προσέγγιση, σφαιρική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα αντίτυπο. Είναι αρκετά ογκώδες, αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Σε 10 λεπτά θα έχουμε την Επιτροπή. Θα έρθουμε, ε, τώρα θα περάσω γρήγορα στο 17 και στο 18 που αφορά τη Συμφωνία Ελευτικής Σύμπραξης με τις Κομόρες. Ο συγητής μας είναι ο Νόρμπερτ. Και νομίζω ότι μας λες ότι θα πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να μας εξηγήσει τώρα γιατί. Sorry, Norbert, said we, move on now to Νομίζω είπαμε ότι πάμε τώρα στο 17 και στο 18 που είναι οι κομμόρες. Θα συζητήσουμε μαζί το 17 και το 18. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για την ε, ε, καταγγελία της ε, Συμφωνίας Σύμπραξης με τις Κομόρες και πιστεύω ότι μη δηλωθήσεις παράνομες και άναρχες πρακτικές αλίες δικαιολογημένα θεωρούνται ότι προκαλούν τεράστιες οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές ζημίες. Αυτή η μορφή αλία συνιστά μια τεράστια απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και έχει σαν συνέπεια η υπεύθυνη αλής πολύ άδικα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και η αγορά της αλίας υπονομεύεται. Η καταπολέμηση αυτής της άναρχης ε, και λαθρέας και παράνομης αλίας είναι ένα βασικό εργαλείο ούτως ώστε να έχουμε μια βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, δυστυχώς είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς προς αυτές τις μορφές αλίας γιατί έχουν μειωμένες δυνατότητες δυνατότητες ελέγχου ε, και επίβλεψης των υδάτων τους. Ε, γι' αυτό γίνονται στόχος αλλιέων που εφαρμόζουν ακριβώς αυτή την παράνομη λαθρέα και άναρχη μορφή αλίας. Ε, μια σειρά διεθνών εργαλείων είναι η βάση για την καταπολέμηση αυτής της μορφής αλίας και φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να κάνει ό,τι μπορεί ε, για να καταπολεμήσει αυτή τη μορφή παράνομης αλίας. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ε, σε μια πληθώρα ψηφισμάτων τονίσει ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση αυτής της μορφής παράνομης αλίας και με το σκεπτικό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέσπισε ένα κανονισμό που αφορά την αντιμετώπιση ε, χωρών που δεν ε, συνεργάζονται και περιλαμβάνει πολλά στάδια μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο διάλογος. Ε, είμαι ικανοποιημένο με την αιτιολόγηση της Επιτροπής έναρξη διαδικασίας για μη συνεργαζόμενες χώρες βάσει αυτού του κανονισμού αλίας και αυτό για πρώτη φορά αφορά τις κομόρες. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα έπρεπε να πούμε ότι επιθυμούμε έναν συνεχιζόμενο πολιτικό διάλογο με τις Κομόρες ούτως ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ε, ε, καθοδήγηση των λευτικών δραστηριοτήτων. Είμαι υπέρ λοιπόν ε, να μην εγκαταλείψουμε την περαιτέρω χρηματοδότηση και ενίσχυση της ε, χώρας. Okay, so, um, anybody... Ωραία. Έχει κάποιες παρατηρήσει λέει, ε, πρόεδρος από αυτού, ο κύριος Σαφχάουζερ. Έχετε το λόγο. Euh, Α, είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε και συμπαθάτε με που ε, δεν ήρθα χθε στη συνεδρίαση, αλλά είχα κάποιο πρόβλημα Πάρα πολύ σωστό είναι να καταγγέλουμε αυτή την αλληλευτική συμφωνία. Το θέμα είναι το πόσο, όπως τόνισε και ο συνάδελφος, οι κομμόρες δεν έχουν τον τρόπο, τα μέσα να μπορέσουν να εποπτεύσουν, να ελέγξουν την ε, αλληλεμπά και γίνεται να συγκροτήσουμε μια επιτροπή εκεί στο Επιτροπή Ειδικού Ωκεανού διότι ήταν μια κάποια λύση Μία λύση είναι οι κυρώσει. Και να δούμε πώς η χώρα μπορεί να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία και να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε τους ωκεανούς και τις ακτές. Όμως αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Κομόρες, ισχύει και για τη Μαυρετανία. Να, οι Γάλλοι είμαστε δεύτεροι στα τις Δεν, δεν, δεν, ούτε εμείς έχουμε τα μέσα να ασκήσουμε τους καταλήλους έλεγχους. Φανταστείτε τι γίνεται στις Κομόρες. Να το πρόβλημα. Πώς να σας το πω. Δεν ωφελεί να καταγγέλει κανείς τα προβλήματα χωρίς να έχει τις απαντήσεις. Ή πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλο να ζητεί το λόγο. Οπότε να δώσουμε το λόγο στην Κατρίνη Σαμπό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την Γενική Διεύθυνση για τη Θαλάσσια Πολιτική. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Η καταγγελία αυτής της ε, συμφωνίας αληφτική σύμπραξης είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το ότι δεν συνεργάζεται για την παρανομιαλία αυτή η χώρα όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Και επενθυμίζω ότι η σχετική διαδικασία της επισήμανσης του προβλήματος με τη χώρα δεν έγινε έτσι στα ξαφνικά, δεν έγινε έτσι αυθαίρετα. Έχουμε πάρα πολλές συνομιλίες πριν αρχίσουμε την προκαταρκτική διαδικασία το 2015 και στη συνέχεια άρχισαν οι επίσημες επαφές και έτσι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείσει τη χώρα να κάνει διόρθωση πορείας. Τώρα, όμως οι κομμόρες δεν τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. και επιτρέπουν την αλληλεία σε διάφορα σκάφη χωρίς να τα ελέγχουν. Οπότε έχουμε παραμελία. Και στις κομόρες και αλλού στους ωκεανούς. Αλλού στον ε, Ανατολικό Ατλαντικό. Άρα, έχουμε εγκαλέσει τη χώρα να συμμορφωθεί. Δεν έκαναν τίποτα. Οπότε και ακολουθούμε την επίσημη διαδικασία της επισήμενης ταυτοποίησης και εμείς πάβουμε την συνεργασία. Άρα, αυτό είναι νέα φάση. Αυτό το διάλογο, το ώστε να μπορέσουμε να αναγκάσουμε τη χώρα να συμμορφωθεί. Επομένως, αυτή η συμφωνία δεν είναι συμφωνία που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά σκάφη να αλλιεύσουν άπαξ και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις βιώσιμης αλίας ε, δεν το κάνουμε αυτό δεν στέλνουμε και τα αλλιευτικά μας γι' αυτό και προχωρήσαμε σε αυτή τη φάση της καταγγελίας και είπαμε ότι έχουμε πρώτα πρώτα το διάστημα της όχλησης που κρατάει ένα εξάμεινο και Εάν θεσπιστεί η κατάλληλη νομοθεσία στη χώρα, τότε θα το πάρουμε πίσω το θέμα της καταγγελίας. «600.000 ευρώ ετησίως είναι ο κύκλος εργασιών της ε, αλία στη χώρα, που στον προπολογισμό της χώρας περίπου αυτό βέβαια. Τέλος πάντων δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά το νεολόγιο και αυτά τα, τα σκάφη αναψυχής ή όχι που αναφέραμε αυτά όσον αφορά την καταγγελία της Συμφωνίας Ελευτικής Σύμπραξης θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι λέει πρόεδρος Κύριος Νόη. Ναι, ίσως εν συντομία, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξή. Από νομική άποψη, δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο δράση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τις κομόρες. Νομίζω ότι νομικά είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τη σύμβαση αυτή, τη συμφωνία αυτή, μετά από μακρές διαβουλεύσεις ε, που δεν βρήκαμε άλλη λύση. Βεβαίω είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε διάλογο με τη χώρα για να, μπορέσουμε να, να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Ναι, υπάρχει αυτή η προθεσμία των έξι μηνών και βέβαια θα συνεχιστεί ο διάλογος. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Είναι 13 του μηνός. Τώρα θα καλέσουμε την Επιτροπή να Συνεχίζουμε δύο σημεία ακόμη. Έχουμε στην ημερήσια διάταξη που είναι επίση πολύ σημαντικά. Και το πρώτο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, ένα από, το, από τα βασικά σημεία της δουλειά μας μέχρι τις ευρωεκλογέ του 2019 και αυτό είναι η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας του Κοτονού μετά το 2020. Έχουμε εκπονήσει έκθεση και στο παρελθόν. Ο Νόρμπερτ Νάουζερ ήταν ε, ο εισηγητής μας. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συστάσεις με απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων και ε, γι' αυτό ακριβώς ήρθε εδώ ο Επίτροπος Μιμίτσα να μας ε, παρουσιάσει σήμερα. Καλή χρονιά, Επίτροπε, ε, γιατί φαίνεται ότι έχει περάσει πολύ καιρό ε, από τις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη φορά που σας βλέπουμε στην Επιτροπή μας με τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά, λοιπόν. Θα θέλαμε να ακούσουμε ποιο είναι το σχέδιά σα για τη Συμφωνία του Κοτονού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πράγματι, καλή χρονιά, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι. Το περασμένο Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση για τη διαπραγμάτευση των οδηγιών για μια απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την συνεργασία των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ μετά από το 2020. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην, στον καθορισμό του μέλλοντος ε, του πιο περιεκτικού, ε, της πιο περιεκτικής και της πιο μεγάλης ε, συνεργασίας στον κόσμο. Πάνω από 100 χώρες, 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι και η πλειοψηφία στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, σε έναν όλο και πιο αλληλοσυνδεόμενο ε, και παγκοσμιούμενο κόσμο αυτές οι σχέσεις είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Είναι η χρονική στιγμή να μεταγράψουμε τη μακροχρόνια στρατηγική μας, ε, συνεργασία μας σε μια πιο στρατηγική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Όπως ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής ε, είπε, ε, θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ ε, την σημασία αυτής της συμφωνίας. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και για το παρόν και για το μέλλον. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πολύτιμη τη δική σας επικοδομητική συνεργασία, τη συμβολή στην επίτευξη αυτών των στόχων και συμπεριλαμβάνω βεβαίως την πρόσφατη έκθεση του κυρίου Νόιζερ. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, τιμώντας τη δέσμευσή μας να σας ε, ενημερώνω πλήρως και να συμμετέχετε πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Η σύστασή μας ήταν αποτέλεσμα διεξοδικών διαβουλεύσεων που έλαβαν υπόψη τα σχόλια και τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα επίπεδα κυρίως ε, από, τις, ε, από τους Ευρωπαίους εταίρους μας αλλά και από τους Αφρικανούς εταίρους, τους εταίρους από τον Ειρηνικό και την Καραϊβική στην ΑΕΤ τον, τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίασα τα πρώτα συμπεράσματα στην κοινή συνεδρίασή μας από κοινού με την ε, ύπατη εκπρόσωπο. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή βάση συζήτησης. Δεδομένη της ε, καλής συνεργασίας μας ε, μέχρι σήμερα, υποθέτω ότι και εσείς θα θεωρήσετε ότι οι προτάσεις μας ε, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Επιτροπής σας. Έχουμε μια φιλόδοξη πρόταση, η οποία ανοίγει το δρόμο για ένα πιο μοντέρνο, ε, μια πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη, πιο πολιτική συνεργασία ε, που ομοιάζει με, τις, ε, με το πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Ελπίζουμε μέσω αυτών των προτάσεων να αντικατοπτρίζουμε καλύτερα τη σημερινή πραγματικότητα και την φιλοδοξία της Ευρώπης να είναι ένας πιο αποτελεσματικός και πιο φιλόδοξος παγκόσμιος παίκτη στον κόσμο, ειδικότερα να αποτελέσει τον ισχυρότερο φορέα ε, αναπτυξιακής πολιτικής ε, επειδή υπάρχει βέβαια και η ε, πολιτική μας, ε, την ευρύτερη πολιτική μας ε, αναπτυξιακή, θεωρούμε ότι οι στόχοι αηφόρου ανάπτυξης πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας, γιατί αυτή η συνεργασία είναι ένα υπόδειγμα της θέλησής μας να πρωτοστατήσουμε στην επίτευξη των στόχων του 2020. Ξέρετε ότι με τις χώρες ΑΚΕ μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική αλλαγή στο πλαίσιο των παγκοσμίων φιλοδοξιών όπου ε, συμβαδίζουν τα συμφέροντά μας στο πλαίσιο για παράδειγμα των ε, διαπραγματεύσεων στο Παρίσι για το κλίμα. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε και να τονίσουμε τον πολιτικό διάλογο σε όλους τους τομείς και για όλους τους στόχους ε, που καλύπτει η νέα συμφωνία. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ε, συγκεκριμένους στόχους, να, να, να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας, της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων, της ασφάλειας, της σταθερότητας, ε, της ε, κινητικότητας και της μετανάστευσης και όπως είπε και όπως αναφέρει και ο κύριος Νόιζερ στην έκθεσή του, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια νέα σχέση ε, εταιρική, ισότιμη, η οποία υπερβαίνει την ανάπτυξη και τον, ε, τον, τις, τις παροχημένες μεθόδους ε, συνεργασίας δικαιούχων και δωρητών. Πολλοί, πολλές χώρες μας, πολλές, πολλοί εταίροι μας είναι πλέον χώρες μέσου εισοδήματος, με διαφορετική διαφορετικά, διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται από τις συμφωνίες συνεργασίας μας και πρέπει να είναι στο καλύτερο, στο πιο κατάλληλο επίπεδο, είτε σε επίπεδο ΑΚΕ, είτε σε επίπεδο περιφερειακό και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβάνωμένων εκπροσώπων των κοινοβουλίων και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ε, τις ε, υψηλές μας φιλοδοξίες και, την, και για την επίτευξη των στόχων μας πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η μελλοντική μας συνεργασία πρέπει να πλαισιώνεται από ένα δεσμευτικό πλαίσιο αυτό είναι βέβαια μια προσέγγιση πολυμερισμού η οποία είναι στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος. Αυτά τα στέρεα θεμέλια θα ε, εκπροσωπούν και τις ε, θεμελιώδεις αξίες μας και θα μας δίνουν την ευελιξία να έχουμε μια πιο στοχοθετημένη αντίδραση ανάλογα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Αυτή η νέα δομή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ε, αυξανόμενη σημασία των περιφερεια, της περιφερειακής δυναμικής και των περιφερειακών φορέων. Πρέπει το κέντρο βάρους δηλαδή να πάει προς τη μεριά των τριών περιφερειακών εταίρων μας που έχουν τις δικές τους κυβερνητικές δομές και τις δικές τους προτεραιότητες περίπτωση της Αφρικής, για παράδειγμα. Ε, η μελλοντική μας σχέση συμφωνία συνεργασίας πρέπει να ενθαρρύνει μια ενιαία προσέγγιση για την Αφρική, ε, λαμβανωμένων υπόψη των συμφωνιών ε, σύνδεσης που έχουμε με τις βορειοαφρικανικές χώρες. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Δεδομένης αυτής της ε, ε, ε, επισκόπησής μου, ελπίζουμε ότι στις βασικές αρχές, ε, στις βασικές κατευθύνσεις συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι πιο σύγχρονη η εταιρική μας σχέση, πιο βασισμένη στην ανταπόκριση ε, υπέρ της προστασίας των κοινών στόχων και των δεσμεύσεών μας ε, και ενίσχυση βέβαια των κοινών μας προτεραιοτήτων και του διαλόγου. Και όσον αφορά την ανάγκη για μια υπεύθυνη και αξιόπιστη Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία με τις χώρες ε, ΑΚΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις ε, διεξοδικά με τα κράτη-μέλη κατά τους ερχόμενους μήνες ε, με στόχο να καταλήξουμε σε μία συμφωνία επί της ε, εντολής την οποία θα έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι το Μάιο. Εγώ βασίζομαι στη δική σας συμμετοχή και στην συνεχή σας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ της ε, δικής σας πρότασης ε, και των όσων ψήφισε η Επιτροπή μας. Όμως, ε, θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος ε, Νόιζερ που ήταν ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Λίντα, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα είπατε. Νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα βασικά σημεία που αναφέρατε. Είπατε ότι είναι μια συμφωνία με μοναδική αξία, ότι πρέπει να καταστεί ε, μια πιο στρατηγική ε, πλατφόρμα και νομίζω ότι έχουμε τώρα αυτή την ευκαιρία. Από τη Βουλγαρική Προεδρία, γιατί εχθές παρουσίασε τις ε, προτεραιότητές της και τις δραστηριότητές της για το επόμενο εξάμεινο και νομίζω ότι είναι ένα προνόμιο το ότι έχουμε με το μέρος μας στην Προεδρία. Θα ε, εμπλακούν πάρα πολύ στη συνέχιση και την παρακολούθηση της Συμφωνίας Κοτονού. Είπατε ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία μας με τις χώρες ΑΚΕ. Προφανώς αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες εντός της συμφωνίας ε, να καταλήξουμε σε ε, πλειοψηφίες στον ΟΗΕ και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε τον πολιτικό ε, διάλογο και Νομίζω ότι εν προκειμένου πρέπει να ε, δεδραματίσουμε το ρόλο μας ως ε, ευρωβουλευτές γιατί είχαμε μια πολύ καλή εμπειρία με την κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση και οι δύο πλευρές πρέπει να βελτιωθούν αλλά αυτό το κοινοβουλευτικό μέσο είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά σημαντικός είναι και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αυτός ο διάλογος νομίζω ότι έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα ως προς τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ε, συνέχιση ε, της ε, Συμφωνίας Κοτονού πρέπει να είναι ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύει τη νέα δομή που σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη για την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό ε, και των βορειοαφρικανικών ε, χωρών βεβαίως ε, θα καλύπτει την Αφρικανική Ένωση γιατί εξ όσων γνωρίζω δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα εντός κάποιων κρατών μελών η διπλή δομή Αφρικανική Ένωση σχέση με την Αφρικανική Ένωση και με τις χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο των χωρών ΑΚΕ το τελευταίο σημείο που θα ήθελα μία ακόμη φορά να τονίσω είναι η συνεργασία με τους ε, βουλευτές και να έχουμε αυτή την καλή εμπειρία. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμφωνία από κοινού με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περισσότερα από αυτά που μας είπατε συνάδουν πλήρως με τις αποφάσεις Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε πολύ, Νόρμπετ, λέει η Πρόεδρος. Ο Άνταμ Σένφελ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ πάρα πολύ θετική τη συζήτησή μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Είναι πολύτιμη αυτή η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια εκτός Ευρώπης. Και δεν μιλώ μόνο για οικονομία και κοινωνία. Μιλώ και για την πολιτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της ε, βοήθειας ούτω ώστε να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα στο μέτωπο αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση τέτοιων στόχων παντού στον κόσμο στόχων πολιτισμού. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις χώρες ΑΚΕ. Εδώ και δεκαετίες έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε αποτελέσματα και επομένως θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι δεν έγινε σωστή στοχοθέτηση. Όμως, αν προκειμένου, επί τόσα χρόνια έχουμε μία δράση μας που δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα, επομένως μπορεί, δεν μπορούμε παρά να νιώσουμε απογοήτευση. Άρα θα πρέπει να γίνει διόρθωση πορείας, όχι επιφανειακή, αλλά εις βάθος. Και γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ θετικά τα όσα μας είπε ο κύριος Επίτροπος που μας μίλησε για το ότι υπάρχει βούληση της ε, τροποποίησης εις βάθος της σχετικής συμφωνίας του 19. Επίσης έχουμε και τον εορτασμό των 100 χρόνων από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα έχουμε τον εορτασμό αυτών προς μήνυμα αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο εκείνο. Οπότε ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών χώρων, αλλά και των διαφορετικών υπήρων. Παρά το ότι σήμερα βλέπουμε να αναδύονται και πάλι κάποιες τάσεις ξενοφοβίας και τα σχετικά. Τώρα όσον αφορά τις ε, χώρες και τις κατευθύνες γραμμές, τους προσανατολισμούς που μας εξηγήσατε, θεωρώ ότι θα πρέπει και εδώ να κάνουμε μια διαφοροποίηση όσον αφορά την προσέγγισή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή προσέγγιση ανά διαφορετική περιοχή δεν μπαίνουν στο ίδιο καλάθι όλες οι χώρες και άλλο Αφρική, άλλο Καραϊβική. Επίσης, για την περίοδο του 2020 θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα. Και συμπαθέμε για το παράδειγμα που θα το αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτού του είδους την ε, αυτοτιμωρία, τις ε, ενοχές που έχουμε. Ε, η ιστορία είναι δεδομένη. Είναι δεδομένες και οι εμπειρίες μας από το παρελθόν. Όλες μας οι τύψεις επομένως, οτι, οτιδήποτε έχουμε κάνει και το μετανιώνουμε. Και μιλώ τώρα για τις χώρες που είχαν απικίες στην άλλη άκρη του κόσμου. Εκείνες οι χώρες ακριβώς λόγω των τύψεων έχουν υπερβολικά ανεκτική στάση. Όμως μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι παραγωγική. Γιατί τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Ε, υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει. Ε, είναι δύσκολα τα πράγματα ιδίω. Εάν ε, δεν, δεν υπάρχουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Γιατί μιλούμε τώρα για κάποιες αρχές πάρα πολύ βασικές, τόσο σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το DNA της Ευρώπης αυτές οι αρχές. είπαμε έχουμε τα χρήματα και θα πετύχουμε τους στόχους, αλλά δεν εξυπηρετείται, δεν, δεν ωφελεί το να εξοδεύουμε χρήματα αν δεν πετυχαίνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Θα πρέπει να αναδείξουμε την ανάγκη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις χώρες μας με τις χώρες εκείνες. Όποιος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου, δεν θα πάρει δεκάρα το ότι χρειάζεστε τη βοήθεια, ε, δεν θα είναι αυτό το καθοριστικό. Άρα, να μην ξεχνούμε ότι σε εκείνες τις χώρες οι κυβερνώντες ωφελούνται από την ε, ενίσχυση και όχι ο κόσμος. Αυτοί που κρατούν τα ενία. Πολλές φορές είναι δικτάτορες. Θα πρέπει όμως να ξέρουν οι εταίροι μας. Εάν δεν πληρούν τι σχετικέ προποθέσει να γίνεται καταγγελία της ε, συμφωνία και να γίνεται ανάκτηση των πόρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει η αρρωγή, η ενίσχυση να μην είναι χωρί προποθέσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς όρισαν βουλευτές από την ε, Γκάμπια και υπάλληλοι του Κοινοβουλίου της χώρας, τους οποίους συναντήσαμε επί μία ώρα την Τρίτη για πρώτη φορά και είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την επιστροφή της δημοκρατίας στην χώρα σας. Μας είπατε τις φιλοδοξίες, τις ελπίδες σας. Ε, πάρα πολύ εντυπωσιακή η ανταλλαγή απόψεων. Ε, θα συζητήσουμε το μέλλον, συζητούμε τέλο πάντων το μέλλον ε, της Κοτονού Μήπως θα ήθελε ο επικεφαλής αντιπροσωπείας να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ να σας τον δώσουμε. Θέλετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ να σας ακούσουμε. So, but we have four more speakers from the Parliament, and if you could bear in mind colleagues to leave time, so we could maybe hear from our, our friends from from from. Um, Έχουμε ζητήσει λόγο και συνάδελφοι, αλλά παρακαλώ να για να αφήσουμε χρόνο για τους συναδέλφους από την Κάμπια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω του συναδέλφου από το Κοινοβούλιο τη Γκάμπιας, καθώ και τον Επίτροπο κ. Μίμητσα, ο οποίο μα ε, παρουσίασε μια αντισύρτηση μετά, στην περίοδο μετά το Κοτονού. Ε, θα πρέπει να επισημάνω δύο σημεία. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια διαφορετική προοπτική από αυτή που γνωρίζουμε εδώ και 20 χρόνια. Σήμερα τα ΙΠΑ αποχωρούν από τις πολυμερείς συμφωνίες, καταγγέλουν και κτημένα στα οποία είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδυναμωθεί από το Brexit. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δύο στοιχεία ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε παραμένει προσυλλομένη στις αρχές του πολυμερισμού, άρα ο ρόλος μας ήταν να γίνουμε πιο ε, να αποκτήσουμε όλο και πιο αναβαθμισμένο ρόλο, έστω και αν ε, οι πόροι ε, παραμένουν ισχνοί. Υπάρχουν χώρες που, στις οποίες επιβάλλονται άλλοι όλοι. Εμείς με μια αρκετά αυστηρή αιρεσιμότητα με το άρθρο 9 πιστεύω το οποίο διαπιστώνει αποκλήσεις σε σχέση με το γραπτό κείμενο και το άρθρο 15 το οποίο προβλέπει κάποιες κυρώσεις. Άρα λοιπόν έχουμε πιο αυστηρούς όρους. Ε, όταν βλέπουμε τώρα στο παρόν πλαίσιο διαπιστώνουμε ότι για άλλες χώρες δεν υπάρχουν οι ίδιοι όροι. Λοιπόν, διαπιστώνουμε επίσης μια αποχώρηση πολλών χωρών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενώ είχαν προσχωρήσει στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, συμφωνίας. 2020. Και η εξέλιξη αυτή είναι σχετική και υπάρχει μια ντουζίνα χώρες που κατορθώνουν να πετύχουν εντυπωσιακέ επιδόσεις. Το ζήτημα των ανισοτήτων βεβαίως δεν είναι αφορά μόνο στις χώρες ΑΚΕ, αλλά υφίσταται επίσης και στην Ευρώπη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Μας είπατε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη, στα νέα δεδομένα. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια... Αναφέρομαι σε κάποια σημεία. Ε, δεν ανέφερα, ξέχασα να πω για την ε, έντονη έντονες δημογραφικές τάσεις στις χώρες ΑΚΕ. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να τις αντιμετωπίσει, να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χωρών και που το επιθυμούν. Γνωρίζουμε ότι όταν εξαγγέλουμε υποσχέσεις ε, είμαστε συσπηρωμένοι, όταν πρέπει να τις εκπληρώσουμε είμαστε 15, 15 η γελία θέση για παράδειγμα παίρνουν κάποιες χώρες σε συζητήσεις που αφορούν ε, το μέλλον των σχέσεών μας ε, με τους άλλους και το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη. Η ερώτησή μου είναι ως εξής. Υπάρχουν χώρες που ανθίστανται στην ε, προσέγγιση ορισμένων θεμάτων στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων. Υπάρχουν ταμπού και αν ναι, και ποιες είναι οι χώρες οι οποίες ε, ε, διαφωνούν ε, στην επίτευξη προόδου σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, η ανταπόκριση στα, στις νέες δημογραφικές τάσεις. Υπάρχουν χώρες που δέχονται να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν και άλλες που αρνούνται να το κάνουν, θεωρούν ότι είναι ταμπού. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε μια στεναρή στάση. Θα πρέπει να έχουμε στους δικούς μας κόλπους μια ανοιχτή συζήτηση. Γιατί έχουμε κάνει κάποιους αγώνες στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε στην πίεση μιας ή δύο χωρών. Θα ήθελα μια απάντηση ειλικρινή. Και κάτι άλλο. Κάποιες παρατηρήσεις που κάνουμε εδώ και ε, κάποια χρόνια. Ε, παρατηρούμε σε ορισμένε περιοχές ε, χωρών ΑΚΕ, ιδιαίτερα σε ορισμένε περιφέρειες, ιδιαίτερα την οικονομική κοινότητα των χωρών της Δυτικής Αφρικής. Εκεί εκπονήσαμε με τη βοήθεια της Επιτροπής ένα σύστημα το οποίο αντιγράφει την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη, διαπιστώνουμε παρόλα αυτά ότι ενώ όλα μας καλούν να υπερβούμε τις αδυναμίες των εθνικών χωρών, ε, η βούληση υπάρχει αλλά δεν είναι αρκετή. Το θέμα της, ένταξης, της ολοκληρής όπως είναι η Τινησία, η Λιβύη, η Αλγερία και το Μαρόκο. Νομίζω ότι το καταλάβατε υπό την έννοια ότι αναφερθήκατε ε, στις πραγματικότητες αυτές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αλλά οι πραγματικότητες αυτές ε, γίνονται όλο και πιο χμηρές ε, η ανθρώπινη εμπορία ε, και άλλα φαινόμενα τα οποία υπερβαίνουν τα εθνικά όρια και αφορούν επίσης ε, ζητήματα σχέσεων μεταξύ Βόρειας Αφρικής, Ποσαχάρης Αφρικής και λοιπά και χωρών και ε, τίποτα δεν είναι εύκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που οι χώρες ΑΚΕ προσπαθούν να αντιγράψουν το δικό τους αναπτυξιακό μοντέλο από την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική αρχιτεκτονική των χωρών αυτών. Η κυρία Χάουτελα, εγώ θα είμαι πολύ συντομότερη από τους προλαλήσαντες, γιατί με περιμένει ένας υπουργός στο γραφείο μου. Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Η ομάδα μας ήθελε να πάμε λίγο πιο πέρα στην ε, αναθεώρηση του εξυγχρονισμού της συμφωνίας. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη περισσότερο τις περιφερειακές ιδιαιτερότητε, αλλά τουλάχιστον εσείς αναφέρατε αυτές τις ε, ιδιαιτερότητε και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν όμως ε, λέτε για το DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ε, αυτή η προσέγγιση, η πολυμερής, πρέπει να πω ότι για το άρθρο 8 δεν ήμασταν πάρα πολύ επιτυχοί στη Συμφωνία του Κοτονού οτιδήποτε έχει να κάνει με, ανθρω... με ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές χώρες ήταν ένα πάρα πολύ επώδυνο, ευαίσθητο και εξοργιστικό ζήτημα για τις χώρες εταίρους μας. Πρέπει να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νομικά δεσμευτική συμφωνία ακόμη και για αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα θα ισχύσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, που τονίζει το ρόλο το, της κοινωνίας των πολιτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πώς μπορούμε όντως να την υποστηρίξουμε και να την ε, βοηθήσουμε να συμμετέχει στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ε, εμείς, πολλοί από εμά συμμετείχαμε στη Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Αμπιτζάν και είδαμε ότι πολλέ φορέ ε, μερικές χώρε ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικέ ω προς το να δεχθούν καν μία δήλωση από την κοινωνία των πολιτών. Είπατε ότι θα υπάρξει μία διαπραγματευτική εντολή μέχρι το Μάιο. Θα είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο και για την Επιτροπή και για την δική μας Επιτροπή αν συμμετέχουμε λίγο περισσότερο στις συζητήσεις για την εντολή. Μου φαίνεται πολύ λογικό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης Λισαβόνας έχει αυτή την αρμοδιότητα ε, μια οριστική γνώμη για τι ε, διεθνεί ε, συμφωνίε. Τελευταία μου παρατήρηση. Έχετε λάβει υπόψη αυτήν την προσέγγιση περισσότερα για περισσότερα, more for more, που στην πολιτική, στη συγκεκριμένη περιοχή ε, έχουμε ε, ακολουθήσει. Μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη ανάπτυξη έτσι. Και συμφωνώ ως προς αυτό με αυτά που είπε ο κύριος Γκόρενς. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σαφχάουζερ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Σύντομος θα είμαι υποστήριξη του πολυμερισμού. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει περισσότερο να βασιζόμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και στο ρόλο των μεγάλων ε, ε, χωρών όταν μιλάμε για πολυπολικότητα ε, πρέπει να σκεφτόμαστε και τη Γαλλία μεν αλλά και τη Ρωσία και την Κίνα η οποία η Ρωσία τώρα έχει βάλει πόδι στην Κεντρική Αφρική κανένας από τους στρατιωτικούς όταν είχε γίνει μετα... μεταβίβαση της εξουσίας ήμουν εκεί κανένας δεν το έλαβε υπόψη είναι αυτό. Επίσης, το ανεπαρκές κράτος, ε, τα Εμμυράτα για παράδειγμα, δεν είναι δημοκρατικός ε, πάρα πολύ καλό, ούτε η Σιγκαπούρη ήταν στο παρελθόν, ούτε και η Κίνα. Όμως ανέπτυξαν τις χώρες τους. Η ανάπτυξη δημιουργεί μία μέσα τάξη και σιγά σιγά δημιουργείται δημοκρατία. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί λοιπόν στις κυρώσεις ε, που ε, πλήττουν περισσότερο τους πληθυσμού και όχι τις κυβερνήσεις που πάντοτε ξεγλιστρούν, έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, η ενίσχυσή μας, η βοήθειά μας δεν λειτουργεί πολύ καλά και το αποτέλεσμα είναι πολύ μέτριο. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνεργασία και επειδή κάποτε ήμουν υπεύθυνο για για τη συνεργασία την αποκεντρωμένη στη Γαλλία, αν δημιουργείται μία οδός, η οποία, ένας, ένας, μια πορεία η οποία δεν οδηγεί σε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη χρηματοδότηση για να δημιουργηθεί ανάπτυξη αν δίνει κάποιο φάρμακα και δεν δίνεται τη δυνατότητα σε κάποιον να, να αγοράσει τα φάρμακα, όλο περισσότερα φάρμακα πρέπει να δίνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό, το ίδιο συμβαίνει και με την αποχέτευση. Ε, τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Το βασικό πρόβλημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε πλούτο σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο εγώ τίποτα δεν έχω να χάσω πια, ε, σε επίπεδο επαγγελματικό ε, επίσης. Ε, προσπάθησα να πω ότι η Κεντρική Αφρική είναι μια χώρα δημοκρατική, υπάρχουν δημοκρατικές εκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός δωρητής. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια λογική ανάπτυξη αποδεικνύει ότι δεν τα καταφέρουμε ποτέ και πάντοτε θα υπάρχει εξάρτηση της, ε, από τη βοήθεια που όλο και περισσότερη βοήθεια ε, ζητά. Λοιπόν, ταμεία Μπεκού, ταμεία ανάπτυξη. καλή πρωτοβουλία είναι αυτή και πρέπει να υποστηριχθεί. Το βασικό σφάλμα, το κύριο σφάλμα και το λέω και το επαναλαμβάνω είναι ότι το κάνουμε εκτός των κρατικών αρχών. Ποτέ δεν θα επιτύχετε την ανάπτυξη μιας χώρας χωρίς κράτος. Οποιοδήποτε κράτος πάρτε, οποιαδήποτε χώρα που αναπτύχθηκε, πάντοτε το κράτος το έκανε. Το να, θέλει να, θέλουμε να υπάρχει ένα μέσο μόνο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή για τις ε, εθνικούς ε, οργανισμούς ανάπτυξης δεν τα κατάφεραν. Για ποιο λόγο θα τα, καθαρίσουν, θα τα καταφέρουν αύριο λόγω ενός νέου Ταμείου Ανάπτυξης. Πρέπει όλα αυτά να πλαισιωθούν από το κράτος και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ μίλησα μαζί του πριν από 10 μέρες για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η δημοσιονομική βοήθεια είναι μια μαύρη τρύπα όπου όλα εξαφανίζονται. Αλλά αν υπάρχει ένα ταμείο ανάπτυξη, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, υπάρχει μια επιτροπή συντονισμού για την υγεία, ε, για τη διατροφή, για την επιτιστική ασφάλεια, ε, για την ασφάλεια της ανάπτυξη αν υπάρχει ένα διπλό κλειδί, ένα κλειδί που έχει η κυβέρνηση και άλλο ένα κλειδί, μιλάω τώρα για υπογραφές, έτσι, για να μπορεί κανείς να... Ε, ε, εκταμιεύει, επειδή έχετε ε, ε, ε, συγκεντρώσει και τους κυβερνητικούς και, με τους, κυβερνητικ... και τους μη κυβερνητικούς φορείς, επιτρέπεται να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα λόγω του συντονισμού και πλαισιώνεται αυτό από το κράτος, γιατί το κράτος έτσι παραμένει το επίκεντρο. Δεν θα υπάρξει ποτέ ανάπτυξη χωρίς την υποστήριξη του κράτους και του πληθυσμού για να υπάρξει, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Σήμερα τα μέσα μας δεν το επιτρέπουν. Πρέπει να αλλάξουμε τα μέσα μας, να τα προσαρμόζουμε. Οι νέες πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να απεμπλακεί η κατάσταση ε, της ε, ανάπτυξης. Εδώ θα συζητήσουμε τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή του δημοσιονομική υποστήριξη γιατί έχουμε ένα ειδικό θέμα γι' αυτό στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα. Ο κύριος Κόγνεγε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε και πάλι στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ήρθα για να μιλήσω για κάτι το οποίο με απασχολεί και με καιρό και πολύ καιρό. Τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα τη αρρωγή, Είναι πολιτικό. Είναι πραγματικό το πρόβλημα. Το θέμα δηλαδή το ότι δεν παρέχουμε, δεν εκταμιεύουμε, δεν πληρώνουμε όσα ε, αναγγέλουμε. Σημαίνει ότι οι χώρες αυτές λένε ότι εμείς έχουμε μπερδέψει τα πράγματα και έτσι δεν ολοκληρώνεται κάθε προσπάθεια. Δεν εκταμιεύονται τα χρήματα τα οποία εξαγγέλλονται. Είναι θέμα προπολογισμού, όχι εισφορά των ε, χώρων. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ούτω ώστε να εκταμιεύονται και να προωθούνται τα χρήματα. Και βέβαια ένας λόγος είναι η Άγγλο-Σαξονική δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οπότε έχουμε 200 περιφέρειες 21 χώρες ε, μόνο γαλλόφωνες οπότε δεν υπάρχει ε, η υποδομή η διοικητική για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που πρέπει αυτό που είπε ο κ. Σαφχάουζερ θα έχουμε στο μέλλον συνέπειες. Άρα θα πρέπει να λάβουμε την πρωτοβουλία ούτως ώστε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων να πάνε στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση των εταίρων μας, ούτως ώστε εκείνοι να μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Και επίσης να βοηθηθούν και αυτοί που υπηρετούν στις αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να έχουμε 100% απορρόφηση των πόρων. Και δεν λέω για τους ε, πολιτικούς, λέω ότι θα πρέπει ή όχι να ε, εκπαιδεύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλου. Και έτσι να είναι πιο ποιοτικέ εκεί οι διοικήσεις. Να ξέρουμε δηλαδή ότι θα πιάσουν τόπο τα χρήματα τα οποία εκταμιεύουν. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήταν ο τελευταίος βουλευτής που έχει ζητήσει το λόγο, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιακούμπα ζετερ τον την αξιότιμη βουλευτή. Για πέστε μας πώς το βλέπετε κατόπιν όσων ακούσατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μας ε, κάλεσε. Πραγματικά ευχαριστούμε όλη η αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης της Γκάμπια. Μέχρι τώρα πολύτιμη αυτή η εμπειρία. Ε, ενημερωθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν επομένως μια ευκαιρία εμείς να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις από διαφορετικές χώρες για τόσα θέματα για τη μετανάστευση, για την αναπτυξιακή βοήθεια και όλα τα άλλα. Πολύ χρήσιμε θα είναι αυτές οι πληροφορίες όταν γυρίσουμε και θα κληθούμε για τα σχετικά να κρίνουμε και να αποφασίσουμε ως βουλευτές. Είμαι η μόνη βουλευτής ε, και ευχαριστώ τους αδέλφους που μου παραχώρησαν την προτεραιότητα να τοποθετηθώ και να μιλήσω. Να σας πω Ποιο είναι το ιστορικό μας πλαίσιο. Πώς καταλήξαμε στην δημοκρατία σήμερα. Έχουμε το άρθρο 9 του Κοτονού, το οποίο άρθρο ορίζει σχετικά και προηγήθηκαν 22 χρόνια δικτατορία στη χώρα μας. Και η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση περιοριζόταν στον πρέσβη ε, και υπήρχαν προβλήματα λόγω της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα. Και αποχώρησε αυτό ο πρόεδρος Πάντως τώρα ως ε, Βουλή πρόσφατα θεσπίσαμε και εγκρίναμε έναν ε, νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Επίσης άλλο νόμο όσον αφορά την Επιτροπή Συμφιλίωσης για να διαχειριστούμε το παρελθόν μας, να πουλωθούν οι πληγές Τη χώρα. Και επίσης συγκροτήσαμε και Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης για ένα νέο σύνταγμα που θα προσφέρει εγγυήσεις για διαίρεση των και διάκριση των εξουσιών και εγγύηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Οπότε ως κυβέρνηση και ως κοινοβούλιο τώρα είμαστε στρατευμένοι υπέρ δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Να δούμε πώς αυτή η νέα μας δημοκρατία να διαρκέσει για πάντα. Τώρα όσον αφορά την ενίσχυση, ο πιο σημαντικός μας εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα, δηλαδή το 2017, όπου τα μια κυβέρνηση, είχαμε αυτή την δημοσιονομική υποστήριξη, είπατε για πηγάδι δίχως πάτο, αλλά μας βοήθησε πραγματικά να ξαναστηθούμε στα πόδια μας. και η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε μία κατεστραμμένη διαλυμένη οικονομία. Και μία στις υποθέσεις σας για να μας δώσετε τη βοήθεια είναι ότι θα έπρεπε να προβούμε σε μεγάλες περικοπές του προπολογισμού. Και για πρώτη φορά στην ιστορία μας καθίσαμε οι βουλευτές και κάναμε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Και λόγω της δημοσιονομικής στήριξης σώθηκε η οικονομία μας. Οπότε δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτή την υποστήριξη. Ξανα ε, στήθηκε η χώρα στα πόδια της. Τώρα, όσον αφορά τη βοήθεια προς χώρες, τη βοήθεια την αναπτυξιακή, ξέρετε χθες είχαμε μια διακοινοβουλευτική συζήτηση και η κάθε χώρα είπε την απόψή της για τη μετανάστευση. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, στη χώρα μας, 99% των μεταναστών είναι νέοι, 15 μέχρι 25 ετών. Και ο λόγος είναι είναι, ο λόγος είναι φυσικά οικονομικός. Όπου υπάρχει βέβαια φτώχεια, ό,τι νόμοι και να ισχύουν, ο κόσμος μεταναστεύει. Οπότε θα πρέπει οι χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί θα πρέπει να αναπτυχθούν γιατί αλλιώς θα συνεχιστεί η μετανάστευση. Και νομίζω ότι η Ευρώπη και η Αφρική θα πρέπει αυτά να τα ατενίσουν με ειλικρίνεια. Αν δεν βοηθά η υποστήριξη για να δείξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα επενδύσεων. Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει όλη την εικόνα της ενίσχυσης και θα είναι ένα αυθεντικό πρόγραμμα επενδύσεων και θα αλλάξει όλη η υπόθεση της ενίσχυσης. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους ε, ενίσχυση που δεν βοηθά. Παίρνουμε λεφτά, ξαναπαίρνουμε, ξαναπαίρνουμε, αλλά δεν βλέπουμε διαφορά. Άρα πρέπει να κάτσουμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο για το πώς αυτή η ενίσχυση θα αποδώσει περισσότερους καρπούς για τις φτωχές χώρες. Εμείς υπολογίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως χώρα δεν έχουμε πολλούς φυσικούς πόρους. Είμαστε βέβαια σε φάση μεταβατική και άρα χρειαζόμαστε βοήθεια για να ορθοποδήσουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Διότι για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο θα κατέβει στο Κοινοβούλιο για έγκριση και θα, αποκτήσει. θα ε, την ε, αναπτυξιακή μας πολιτική. Έχουμε πέντε προτεραιότητες. Υγεία, χειραφέτηση των νέων, παιδεία, γεωργία και υποδομές. Είναι οι πέντε προτεραιότητες της χώρας. Οπότε κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη. Ξέρετε, κάναμε περικοπές 200 εκατομμυρίων από άλλα κεφάλαια του προβλησμού να τα πάμε στο κεφάλαιο της υγείας γιατί το σύστημα υγείας καταραίει. Επομένως, κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη και πάλι σας ευχαριστούμε μας δίνει ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ με την πρακτική σας εμπειρία, γιατί εδώ μιλάνε οι συνάδελφοι για την δημοσιονομική στήριξη, κατά πόσο δουλεύει ή όχι. Εσάς ε, ε, σε εσά ε, λειτουργήσε. Μας μιλήσατε για τα προβλήματα που είχατε σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν επίση τα ζητήματα πρέπει να υπάρχει κάποια αιρεσιμότητα, γιατί το είπε προηγουμένω ο συνάδελφο. Είπατε ότι υπήρχε, ε, υπήρχαν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο, στη χώρα σας ε, ε και είχαν ε, ανασταλεί τα αναπτυξιακά προγράμματα οπότε συμβαίνει αυτό τώρα όμως έχει επιστρέψει η δημοκρατία και έχουν επανέλθει όλα είναι εδώ ο Επίτροπος παρουσιάζει το ε, σχέδιο διαπραγματευτική εντολής ε, για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας του Κοτονού που θα ε, την παρουσιάσει και σε εμά και στους υπουργού. και εμείς προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε αυτού του είδου στον έλεγχο συζητούσαμε την άλλη φορά. Να δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και για τη συμβολή σας αλλά και για την καθοδήγησή σας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε ένα πολύ, ε, ένας πολύ βασικός εταίρος ε, κατά τις διαπραγματεύσεις ε, και κατά τον καθορισμό της τελικής διαπραγματευτικής εντολής αλλά και στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ε, της ε, συμφωνίας μετά τη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού. Όντως το Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαπραγματεύσει, να διαπραγματήσει, συγγνώμη, με τη σύμφωνη γνώμη του σε σχέση με τη συμφωνία. Δεν θα ήθελα όμως εγώ να έρθω τέλη 2019 στο Κοινοβούλιο με μη, ένα ε, οριστικό κείμενο της συμφωνίας ε, θα ήθελα να ε, συζητώ μαζί σας πιο συχνά, να έρχομαι στην Επιτροπή σας και στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να μπορέσω να ε, ε, ε, λάβω αυτή την υποστήριξη και αυτή την καθοδήγηση που για μένα είναι πολύ σημαντικές. Συμφωνώ απολύτως ότι σήμερα υπάρχει μια διαφορετική προοπτική προκειμένου να δημιουργηθεί το σωστό πολιτικό και αναπτυξιακό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών και για την περίοδο μετά το 2020. Έχουμε τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης, έχουμε τους δικούς μας ε, στόχους, ε, ε, τη δική μας παγκόσμια στρατηγική και όλα αυτά τα έγγραφα για πρώτη φορά άρουν αυτά τα ε, ε, όρια μεταξύ ε, δικαιούχων, μάλλον αυτές τις διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων και των δωρητών είναι στόχοι που αφορούν όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Το νέο μας πλαίσιο με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να αντανακλά αυτές τις νέες προοπτικές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, αντανακλάνε, να αντανακλάτε ε, στο ε, μεγαλύτερο τμήμα της ε, συμφωνίας και ε, στο κομμάτι το περιφερειακό που θα αντανακλά όλες τις ιδιαιτερότητες της μελλοντική συμφωνίας. Αυτή λοιπόν είναι η δομή που προτείνουμε. Μία δομή η οποία ε, θα περιλαμβάνει ένα κομμάτι που αφορά το κεκτημένο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοτονού, τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ε, που, που ε, σκοπό έχει να ε, διατηρήσει τις ε, κοινέ μας αξίες, το κράτος δικαίου, την καλή διακυβέρνηση, την προσέγγιση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά τα κεκτημένα τα οποία ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού και δεν βλέπω κανέναν ε, καλό λόγο να ε, τα εγκαταλείψουμε και να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διαφορετική ή αόριστη ε, συμφωνία που θα είναι λιγότερο δεσμευτική. Και προτείνουμε επίσης τρία τρεις ε, ειδικούς πυλώνες που αντανακλούν την ε, αναπτυξιακή πραγματικότητα και τις αναπτυξιακές ανάγκες του άξονες ανάπτυξης ε, για τις τρεις περιφέρειες συγκεκριμένα. Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός. Συμφωνώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αναβαθμίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο ο οποίος σε διμερές επίπεδο με τις χώρες εταίρους αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου υπό το άρθρο 8 ε, της ε, ισχύουσας συμφωνίας του Κοτονού είναι ένα σημαντικό εργαλείο είναι ένας ε, σημαντικός ε, μοχλός για να μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε, να διατηρήσουμε αυτά τα σημαντικά σημεία που στοιχειοθετούν την προσέγγισή μας από τη μία λοιπόν πρέπει να αναβαθμίσουμε τον πολιτικό μας διάλογο από την άλλη πρέπει να κάνουμε τη διάκριση σε σχέση με το άρθρο 96 της τωρινής συμφωνίας που αφορά την αναστολή αυτή τη στιγμή ο πολιτικός διάλογος δεν οδηγεί ε, πλέον σε ε, καλό αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει μια διάκριση σαφής μεταξύ του πολιτικού διαλόγου και του άρθρου 96 και πρέπει να συμφωνήσουμε, μεταξύ, να συμφωνήσουμε για τις ε, ειδικέ κυρώσεις, αναστολές και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια αιρεσιμότητα μεταξύ μιας προσέγγισης βασιζόμενη στα δικαιώματα και των αναπτυξιακών προγραμμάτων ε, στην νέα συμφωνία που θα υπάρξει να έχουμε ένα πλαίσιο δηλαδή που θα ορίζει καλύτερα αυτή την προσέγγιση more for more, ε, περισσότερα για περισσότερα, η οποία στρατηγική βέβαια, η οποία προσέγγιση θα ορίζεται καλύτερα ακόμη στο πλαίσιο των περιφερειακών ποινών που ανέφερα προηγουμένως. Οπότε για τους ερχόμενους μήνες, ελπίζω ότι οι ερχόμενοι μήνες θα είναι μόνο και ότι δεν θα πάρει πολύ περισσότερο, τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν μέχρι το Μάιο για τη διαπραγματευτική εντολή και μετά να αρχίσουμε ε, το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Το είπα πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Για δεν θα πρέπει να είναι η καθαρά παραδοσιακή ε, διαπραγμάτευση. Ε, πρέπει να είναι περισσότερο ένας συνεχής διάλογος μεταξύ των εταίρων πώς μπορούμε να θέσουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο, σύγχρονο πλαίσιο για το μέλλον, μια πολιτική και οικονομική αναπτυξιακή σχέση. Αυτό νομίζω ότι διακυβεύεται εδώ και σε αυτό βασίζομαι στη δική σας συνεισφορά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Επίσης, να συμφωνήσω με όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές ε, που χαιρέτησαν ε, την παρουσία και τη συμμετοχή των συναδέλφων μας από το Κοινοβούλιο της ε, ε, Γκάμπιας. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μπορούμε να επανεπισημάνουμε ε, και πάλι την την υποστήριξή μας στην χώρα σας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της χώρας σας ε, στην ε, μελλοντική συμφωνία, στο πλαίσιο που θα υπάρξει μετά το πέρα συμφωνίας του Κότονου. Εμείς πραγματικά περιμένουμε τη συμμετοχή σας ε, και ελπίζουμε ότι θα μπουν σε μια σωστή κοινή πορεία, σε μια πορεία εταιρική σχέσης πολλά θέματα για την οικονομική ανάπτυξη, για τη διαχείριση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης, των μεταναστευτικών ροών. Η Γκάμπια βρίσκεται σε μία ε, κρίσιμη καμπή μετά από 22 χρόνια ολοκληρωτισμού. Οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις είναι τεράστιες. Ε, μετανάστευση, ε, ενέργεια, ασφάλεια. Νομίζω όμως ότι η προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους και η περιεκτική ανάπτυξη βεβαίως, χωρίς αποκλεισμούς δηλαδή, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ευημερία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να συνοδεύσει τις εθνικές ε, αναπτυξιακές προτεραιότητες. Εγώ ήμουν ο πρώτος ξένος επισκέπτης ε, που επισήμως ε, επισκέφθηκε την Γκάμπια κατά τη δεύτερη εβδομάδα της ανάληψης καθηκόντων του νέου σας Προέδρου και είχα την ευκαιρία συνεπώς να επανεπισημάνω την πολιτική και αναπτυξιακή μας υποστήριξη ε, για να ε, μπορούν να προοδεύσουν τα αναπτυξιακά μας προγράμματα και θέλουμε κυρίως να σας υποστηρίξουμε ως προς τα μέσα ενίσχυσης οικονομικής ανάπτυξης μέσω δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Ήμασταν εκεί το 2017 μέχρι το 2020 πάνω από 325 εκατομμύρια ευρώ ε, στοιχίζουν τα προγράμματα που είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τον εθνικό διμερή ε, με την εθνική διμερή μας ε, με την εθνική διμερή ε, συμφωνία Υπήρξε λοιπόν δημοσιονομική υποστήριξη αρκετά σημαντική προς την Κάμπια και πραγματικά αναμένω ε, την συνεργασία με τις ε, αρχές της χώρας σας. Ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε και άλλους δωρητές να συμμετάσχουν και, να συμμετάσχουν και εκείνοι σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Θέλουμε να οργανώσουμε μια νέα διάσκεψη δωρητών για την Κάμπια τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Οπότε πραγματικά επικροτώ τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά σας προς την υποστήριξη αυτής της νέας ε, δημοκρατικής ε, εξέλιξης του ανοίγματο της χώρας σας για να μπορέσετε να επιτύχετε όλους τους στόχους ε, που είναι τμήμα του θεματολογίου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας ε, ε, κάνατε αυτήν την ενημέρωση για την Γκάμπια. Βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας από την ε, Γκάμπια και συμφωνήσαμε χθες τους συντονιστές να να δεσμευτούμε για το Κοτονού πριν από τον Μάιο. Ε, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε. Ξέρω ότι είστε τακτικός επισκέπτης στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 20 την ε, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη του προϋπολογισμού με τον Στεβάν Μαντσεβίση, τον ε, διευθυντή της ε, ΔΕΦΚΟ. Σήπαν πόσο σημαντικό είναι από την αντιπροσωπεία της κάπια να τους ε, υποστηρίξουμε και πώς ε, θα πρέπει να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή ε, με ένα πολύ διαφανή τρόπο με την υποστήριξη του προπολογισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό σήμερα το πρωί ακούσαμε μια παρουσίαση για τη ILO για το θέμα της κοινωνικής προστασίας. Και εδώ βεβαίως η υποστήριξη του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική στον αφορά την ανάπτυξη των ε, σχημάτων, των μοντέλων κοινωνικής προστασίας και η Προσπία της Γκάμπια είπαν ότι μοντέλα απασχόλησης και σχήματα κοινωνικής προστασίας ε, θα δώσουν στους νέους ανθρώπους ε, ελπίδα και θα τους στηρίξουν να οικοδομίζουν την δική τους χώρα. Εγώ θα φύγω στη μέση αυτής της ε, παρουσίασης. Αυτό δεν έχει να κάνει με την σπουδαιότητα του θέματος, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αλλά θα πρέπει να συμμετάσχω στον εορτασμό για την επέτειο των 100 ετών από την ε, χορήγηση του δικαιώματος ψηφοφορίας, ε, ψήφου στις ε, γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Στεφάνο έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ Λίντα, σε ευχαριστώ πολύ και πράγματι ακούγοντας την αντιπροσωπεία της Κάμπια σχηματίζει κανείς μια θετική εικόνα γιατί είπαν ε, σαφώς ότι είναι κομμάτι της οικοδόμησης της χώρας τους. Άρα λοιπόν είναι μια καλή εισαγωγή αυτή τη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση η οποία είναι σημείο ε, κίνηση για τη συζήτηση. Τώρα, καταρχήν, η πρώτη διαφάνεια, με κάποιες ε, βοηθητικές διαφάνειες. Έχουμε 13 ε, δις ε, χαρτοφυλάκιο. Έχουμε 265 συμβόλαια υποστήριξη των προπολογισμών, 90 χώρες και συμπεριλαμβάνουν εδώ την, και τη δική μας γειτονία. Βλέπουμε εδώ στην ε, διαφάνεια ε, ποια είναι η διασπορά. Βλέπουμε τις γειτονικές χώρες, ε, νότια και ανατολικά, αλλά και η Αφρική, η Ανατολική και Νότιος Αφρική κλπ. Τα βλέπετε στην διαφάνεια. Άρα λοιπόν δαπανούμε περίπου το 20% στην ε, υποστήριξη του προπολογισμού, 40% μελώντας για τα διμερή προγράμματα. Αν δούμε το σύνολο των ε, δαπανών σε διμερές περιφερειακό επίπεδο κλπ. Ε, υπάρχει μια μείωση τουλάχιστον του 20% αλλά εδώ γεωγραφικά μπορούμε να παρέμβουμε και να σταθμίσουμε τις δαπάνες υποστήριξης του προϋπολογισμού. Και πάλι κάποια αριθμοί ε, έχουμε τρεις τύπους ε, συμβολέων τα συμβόλαια του τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης το δεύτερο είναι το συμβόλαιο παθοτικότητας Στομακής μεταρρύθμισης και, ένα, και η τρίτη κατηγορία, η οποία είναι πιο πρόσφαση, αφορά την οικοδόμηση ανθεκτικότητα στη χώρα, όπως η Γκάμπια για παράδειγμα, όπου ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τη χώρα στην οικοδόμηση. Ε, ε, είναι και το πιο δύσκολο αλλά ε, εδώ υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να έχουμε και μια πολιτική επιρροή. Δείτε τι γίνεται στο Αφγανιστάν και μπορούμε να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά με άλλα μέσα. Και βλέπετε από τη διαφάνεια ότι η αποδοτικότητα της τομεακής μεταρρύθμισης είναι πιο σημαντική γιατί καλύπτει το 83% του προϋπολογισμού μας. Τώρα, εάν ε, σας δώσω τώρα τα στοιχεία, την ε, αποδοτικότητα, γιατί ε, ε, καταβάλω τα χρήματα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Γιατί καμιά φορά στα παρελθόν ήταν ε, ιδέα ότι βάζουμε χρήματα στον προπολογισμό και μετά που τον είδε, που τον ξέρει κλπ. Ε, τώρα όμω ε, τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Βεβαίω μπορούν να υπάρχουν αποτυχίε ή επιτυχίε αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται η προσμέτρηση της επιτυχίας γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα και υπάρχουν τέσσερις ε, γενικοί όροι που θα πρέπει να τηρούν οι χώρες για να μπουν στο παιχνίδι της υποστήριξης του προϋπολογισμού. Μια ε, αξιόπιστη ε, πολιτική, ε, πολιτικ, μακροοικονομική ε, πολιτική που να προσανατολίσει σταθερότητα, ε, μία πρόοδο στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, των δημοσιονομικών και μία διαφάνεια στον προπολογισμό. Το απλό δεδομένο ότι γίνεται διαπραγμάτευση ενός περιεχομένου προπολογισμού πάντοτε συνεπάγεται μία συζήτηση για μεταρρυθμίσεις, για μεταρρυθμίσεις συγγνώμη, για ανοικοδόμηση εφόσον είναι τρωτή η κατάσταση ή μπορείτε να το ονομάσετε βελτίωση της διαχείρισης ή καταπολέμηση της ε, διαφθεράς εξυγένση κάποτε ε, ανάλογα με το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να φέρω σε σχέση με την αποδοτικότητα. Και αν δείτε τη διαφάνεια εδώ, βλέπετε ότι εφόσον συνδυάζουμε το σημείο εισόδου με τη καταβολή της βασικής ε, δόσης, ε, και στη συνέχεια το 50% περίπου της συνέχισης της καταβολής συνδέεται με την αποδοτικότητα και τη συμφωνία με τους πεσυμφωνημένους ε, δίκτες. Εάν ε, ε, και μπορούμε να δούμε τι είναι οι δείκτες για την καταβολή των δόσεων. Για παράδειγμα, νέος νόμος για τις προμήθειες, η εισαγωγή της πληροφορικής, η βελτίωση της ε, διοίκησης ε, της ε, και βεβαίως όλα αυτά αφορούν την διαφάνεια. όταν η κυβέρνηση βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου ή άλλων πολιτικών οργάνων προκειμένου να αποκαλύψει κάποια στοιχεία. Και το output ε, όταν πρόκειται για τομεακές ε, μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα στο τομέα της εκπαίδευσης ή της υγείας, μπορούμε να το προσμετρήσουμε πόσα σχολεία έχουν φτιαχτεί ε, τι γίνεται με τις υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων ή προγράμματα εμβολιασμού ή μητρό καταχώρησης ε, ανάπτυξη στοιχεία. Γιατί, για παράδειγμα, σε ορισμένε περιπτώσει όπω είναι η προγραμματα εμβολιασμου η μητρο καταχωρηση επιχειρησεων η αυξηση της λογοδοσιας ολα αυτα ειναι διακόπτουμε την καταβολή. το ζήτημα της ε, φορολόγησης. Γιατί βεβαίω η υποστήριξη του προπολογισμού συνδέεται με την ε, κινητοποίηση του εθνικού προπολογισμού. Και αφορά την πρόσβαση βεβαίω στις βασικές υπηρεσίες στην προηγούμενη διαφάνεια όπου είδαμε τις γενικές προϋποθέσεις για να είμαστε ξεκάθαροι εφόσον ε, η μία από αυτές τις προϋποθέσεις ε, δεν ε, εκπληρώνεται δεν δίδεται υποστήριξη. Θα πρέπει να εκπληρώνονται λοιπόν και οι τέσσερις. Είναι βασική προϋπόθεση εισόδου στο πρόγραμμα. Εάν δεν, γίνον, δεν τηρούνται οι δείκτες, δεν εκταμιεύονται οι δόσεις. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν πλήρης συμμόρφωση ή, παίζουμε, ή καταβάλουμε ένα μειωμένο ποσό εφόσον πληρούνται εν μέρη προϋποθέσεις. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει και η έκταση δίνει περισσότερα στοιχεία εδώ ότι είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο υποστηρίζει την πολιτική διαλόγου και την ε, αύξηση διαφάνειας ε, όσον αφορά τη συμφωνία των εξαγγελιών της εν λόγω κυβέρνησης με, με την πράξη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μετράμε τις μεταρρυθμίσεις, το output, Ε, και όπως σας είπα καταβάλλεται αρχικά το 50% εάν δεν υπάρχει περαιτέρω συμφωνία είτε καταβάλλεται μια μένη δόση είτε κόβεται εντελώς η χρηματοδότηση. Ε, Τώρα, το κατά πόσο παράγονται συγκεκριμένα αποτελέσματα από το εργαλείο προωθεί τις προσπάθειες εφαρμογής όσον αφορά την ε, μακροοικονομική ε, δημοσιονομική διαχείριση υποστηρίζοντας το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων και εν γέννη τις επενδύσεις σαν ένα εργαλείο συμβολής και βλέπουμε πώς, ε, τώρα εξετάζουμε κατά πόσο μπορούμε να συνδέσουμε πιο συγκεκριμένα το εργαλείο αυτό υποστήριξη του προπολογισμού με την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Γιατί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι ένα μείγμα βεβαίως ε, νομοθετικών αποφάσεων, διοικητικής ε, ικανότητας κλπ κατά πόσο δηλαδή η χώρα έχει την υποδομή για να δεχτεί τις ε, επενδύσεις. Τώρα κάποια άλλα σημεία τα οποία αφορά η διαφάνεια αυτή η ευθυγράμμιση της χώρας με το εθνικό πρόγραμμα αυτό είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό εμείς ε, παρεμβαίνουμε στον κύκλο προϋπολογισμού που αφορά την πολιτική που έχει αποφασίσει η χώρα σε σχέση βέβαια με τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα δυνατόν να αποβλέπουμε σε ένα μέγιστο βαθμό κυριότητας εκ μέρους της χώρας και μείωση του διοικητικού άχθους. Ε, κόστους. Ενδεχομένως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες αυτές ε, βασίζονται στον πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα ε, εφόσον ανοιχνεύονται λύματα από την πλευρά της χώρας. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί έχει να κάνει με το πόσο εσωτερικεύει αυτή η χώρα τις ευθύνες της. Τώρα άλλη διαφάνεια. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι μηχανιστική η σχέση μεταξύ της δημοσιονομικής στήριξης και του αποτελέσματος. Πρόκειται για κάτι το οποίο στηρίζεται σε στοιχεία, σε ενδείξεις. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται όσον αφορά την ε, φτώχεια. Βλέπετε την, το, πορτοκαλί γραμμή στο γράφημα που αφορά τις χώρες που έχουν στήριξη και όχι οι άλλες. Οπότε βλέπουμε ότι όπου υπάρχει στήριξη έχουμε πιο σταθερή συρρήγνωση του φαινομένου. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί η φτώχεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο. Αφορά δουλειά όλης της χώρας και της ε, κοινωνίας. Να, το πρώτο στοιχείο που θέλω να σας ε, αναδείξω και έχει σχέση με τα στατιστικά. Παρακάτω τώρα. Παιδική θνησιμότητα. SDG 2. Βλέπετε εδώ τις χώρες όπου οι ενδείξεις τονίζουν το ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και βλέπουμε το ότι έχουμε τομεακή στήριξη. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε σημαντική συρρήγνωση του φαινομένου της παιδικής θνησιμότητας. Παρακάτω. Υγιεινή και νερό. Πρόσβαση σε πόσιμο επίσης. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει σημασία ανάληψη δράσης από την χώρα που είναι ο εταίρος μας ό,τι και να κάνουμε εμείς. Αλλά δεν έχουν τις κατάλληλες πολιτικές οι ίδιοι οι άνθρωποι στη χώρα, εκείνα δεν κάνουν τις κατάλληλες επιλογές, δεν γίνεται τίποτα. We can see in terms of, uh, in Burkina Faso, for example, in, in... βλέπουμε δώσουμε την Burkina Faso, τι γίνεται όσον αφορά την περίοδο 2009-2016, να Φάσο, μετά έχουμε την Βολιβία, βλέπουμε ότι ένα και έχουμε αύξηση της πρόσβασης. παρακαλώ τώρα. Έχει σχέση με τη διαχείριση των δημοσιονομικών. Αυτό το είπαμε και στην αρχή, αλλά έχει σημασία αυτό να καταγραφεί, να δούμε, για να είναι κανείς επιλέξιμος τι προϋποθέσεις χρειάζονται. και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν πάλι ενδείξεις βελτιώσεων. Έχουμε εδώ μια σειρά κριτηρίων αξιοπιστία του προϋπολογισμού, κατάρτιση προϋπολογισμού αναπολιτική, έλεγχος δημοσιονομικός. Οπότε εδώ είναι πιο έντονη η βελτίωση, διότι έχουμε μέτρα ελέγχου απλουράς του κράτους. Πολύ σημαντικά αυτά. Και έχουν σχέση με τους ε, στόχους του 16 και 17. Τώρα υπάρχει το θέμα της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Βεβαίως και πρόκειται για έναν κίνδυνο, πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο ελκύει την προσοχή μας. Γιατί ακόμα και έχουμε κάποια μέτρα μείωση της διαφθοράς, αν ό, και όλα γίνουν όπως τα είπαμε πριν, πάλι υπάρχει ο κίνδυνος. Και όλα αυτά στηρίζονται στην εμπειρία μας, η κατανόηση της διαφθοράς έχει αναβαθμιστεί λόγω της δημοσιονομικής βοήθειας. Δεν λέμε ότι υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού και κάποιο είδους αυτοματισμός, αλλά είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του δίκτυ συνειδητοποίησης της ε, διαφθοράς από τον φορέα Transparency International και από την άλλη μεριά τον ε, δίκτυ που προέρχεται από το World governance και βλέπουμε ότι όταν έχουμε δημιουργηθεί στήριξη τότε η κατάσταση είναι καλύτερη όσον αφορά το πόσο αισθητό είναι το φαινόμενο, τη συνειδητοποίηση του φαινομένου. Άρα όταν υπάρχουν συνθήκες κατά τι οποίε οι εμπλεκόμενοι και οι πολίτες εσωτερικεύουν, συνειδητοποιούν το φαινόμενο. Άρα δημιουργείται δυναμική στη χώρα για να αντιμετωπιστεί το δεινό αυτό. Επίσης Έχουμε αυτή την ανάλυση που στηρίζεται σε κάποια στοιχεία και επισυνδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σχετική μείωση της διαφθοράς. Άρα, βελτίωση. Άρα και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Άρα όλα τέλεια, ε όχι βέβαια. θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες επιλογές. Κάθε μήνα θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έχουμε τη σχετική συνάντηση κάθε μήνα. Μαζευόμαστε όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Λέξτε υπηρεσίες εξωτερικής δράσης, ντεύκο Και θα πρέπει να αποφασίσουμε για τον έλεγχο. Πρέπει να αποφασίσουμε για την επιλεξιμότητα να αποφασίσουμε για την ανάλυση του κινδύνου και να αποφασίσουμε τι θα εκταμιευθεί. Και βέβαια οι συζητήσεις αυτές είναι πολύ ζωηρές, διότι δεν είναι πάντα τα πράγματα εύκολα και ομόφωνα. Ας πούμε συνέχεια μπαίνει το επιχείρημα της ισότητας των φύλων. Θα μπορούσαμε σε εκείνη τη συνάντηση τη μηνία να έχουμε και μερικούς από εσά για να δείτε τι γίνεται. Πάντοτε η άμεση συμμετοχή θεωρώ ότι είναι σημαντική. Και όχι να παρακολουθείτε, αλλά και να κάνετε προτάσεις, να συμμετέχετε. Γενικά πάντως είναι success story αυτή μας η προσπάθεια. Θα πρέπει επίσης να ε, επικαιροποιήσουμε τις καθηγητές γραμμές του 17 συνένεση ε, θα πρέπει οι τρεις συμβάσεις να είναι πιο κατανοητές και άρα θα πρέπει αλλιώς να τις ονομάσουμε Links Sectorial Reform State Building και έτσι να δούμε τι θα γίνει με το εσωτερικό εισόδημα επί τη βάση της προσπάθειας για ανθεκτικότητα, για το κλίμα ισότητα των φύλων. Έλεγχος επίσης και να δούμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, ο διάλογος για τις πολιτικές είναι πάρα πολύ ε, δύσκολος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όση γνώση θα οφείλαμε. Είμαστε σε επαφή όσες αντιπροσωπίες και για τον έλεγχο και για την ποιότητα του τομεακού διαλόγου. Πάνω κάτω αυτά περιέχει η έκθεση. Αυτά πάνω κάτω. Ήθελα να ξέρετε για να έχετε τουλάχιστον μία εικόνα του τοπίου. Και μετά τα κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να πάρετε το λόγο. Και θα έχουμε και κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, ε, αν έχει την καλοσύνη, ο κύριος Μανσιβησή να μας απαντήσει. Κύριε Ρούμπικ. Äh, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ε, παρουσίαση. Για μας η παρουσίαση βεβαίως είναι πολύ σημαντική γιατί στη βάση των αποτελεσμάτων του έτους 2017 καταρτίζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή θα πρέπει να δούμε πώς θα επανοριστούν ε, οι προτεραιότητες. Και θεωρώ σημαντικό το ερώτημα που είναι πού έγκυται το βασικό μας καθήκον ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πού θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα πρέπει να βρούμε κάποιους εταίρους να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσεις για να μπορέσουμε να δημορφώσουμε καλύτερα την βοήθεια. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης, όλοι γνωρίζουμε ότι το στοιχείο υπαριθμών 2 είναι το στοιχειώδες, η γεωργία και η γης ε, διατροφή. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καθοριστικά σημεία στην Ευρώπη και τι δυνατότητες έχουμε στον τομέα αυτό. Βεβαίως αυτός ε, εξαρτάται από το πώς ε, θα ελοπίσουμε τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης 7 ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στις ε, περιφέρειες της υπαίθρου ή πώς μπορούμε να επενδύσουμε στον τομέα αυτό τους ώστε να έχουμε βιώσιμη ενέργεια και επίση το σημείο υπαριθμών 6, δηλαδή υγειονομικέ εγκαταστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, είναι πολύ σημαντική η καθαριότητα των, ε, το καθαρό νερό ε, και θα πρέπει να κάνουμε μια ιεράρχηση των επενδύσεων που έχουμε παραδείγματα βέλτιστων τεχνητών στον, στην ενέργεια, στον, στις, ενεργειακές, στις υγειονομικές υποδομές κλπ. Ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνουμε ε, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε και τη χρηματοδότηση που αφορά χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας βεβαίως και είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να φροντίσουμε στις επενδύσεις να είναι καθαρή η προκήρυξη διαγωνισμών, να γίνεται με το σωστό τρόπο και αυτό αφορά και τις εγκαταστάσεις ε, ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας ε, για παράδειγμα, τις επενδύσεις σε τέτοιου είδους έργα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι να το κατοχυρώσουμε και για τις επόμενες γενιές να υπάρχει μια καθαρότητα στις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόιζερ έχει το λόγο. Äh, Ευχαριστώ πολύ και από τη δική μου πλευρά. Πιστεύω ότι ήταν ε, σημαντικό και πάλι να δούμε τι γίνεται με το εργαλείο της δημοσιονομικής υποστήριξης γιατί στην Επιτροπή Ανάπτυξης πάντοτε ε, καλούμε επειδή υπάρχει μια σχετική ζήτηση, το πώς θα χειριστούμε τα χρήματά μας και να δούμε κατά πόσο δεν είναι μεγάλο ρίσκο να στηρίζουμε κυβερνήσεις με άμεση δημοσιονομική στήριξη. Νομίζω ότι στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης ε, στην, με την αντιπροσωπεία της Γκάμπια ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η δημοσιονομική στήριξη για τη χώρα της ιδιαίτερα μετά την κυβερνητική αλλαγή και είδαμε ένα πολύ θετικό παράδειγμα της δημοσιονομικής στήριξης. Αλλά βεβαίως ε, μπορούν να υπάρξουν και περιπτώσεις ε, κακο... Ε, κατάχρησης, κακοδιαχείρισης κλπ. Για παράδειγμα στην ΑΕΤ όπου εκεί είχαμε πάει με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα και βεβαίως ε, εναπόκειται σε εμά να μεριμνήσουμε για την ε, αξιοποίηση των χρημάτων αυτών. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν και οι μηχανισμοί ελέγχου και παράλληλα με τη δική μας Επιτροπή, βεβαίως και η Επιτροπή Προπολογισμών διαδραματίζει εδώ καθοριστικό ρόλο προκειμένου να ελέγξει το πώς ε, δαπανώνουν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. και πώς εφαρμόζονται τα προγράμματα. Ευχαριστώ και πάλι. θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα συμπέρασμα, μια διαπίστωση και μια ερώτηση. Η διαπίστωση είναι η εξής. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε πεπισμένοι ότι η δημοσιονομική υποστήριξη είναι κάτι καλό, έχει αποτέλεσμα θετικό και είχατε την ευκαιρία να το δείξετε κι εσείς. Κατά τη γνώμη μου είναι και μία, ένα τελευταίο στάδιο της απεικιοκρατίας. Δεν πρέπει εμείς πια να λέμε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά η ίδια κυβέρνηση στο βαθμό του δυνατού ε, όταν ελέγχεται από ε, έναν ε, λαό που τον ψηφίζει ελεύθερα και δημοκρατικά να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος για να καταλάβω απλώς, λέτε ότι μία από τις τέσσερις προϋποθέσεις για να είναι κανείς δικαιούχος της δημοσιονομικής υποστήριξης είναι η μακροοικονομική σταθερότητα. Εσείς κάνετε αυτήν την διαπίστωση. Η κυβέρνηση ή το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ που είναι παρόν σε όλες τις χώρες και έχει τις ε, κεραίες του συντονισμένες παντού. Υπάρχει διπλή κάλυψη ή εν πάση περίπτωση υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ των διεθνών φορέων. Ποια στοιχεία έχετε ε, στη διάθεσή σας για να ε, καταδείξετε μια κατάσταση και να αποφασίσετε αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τα στοιχεία του ΔΝΤ να υπενθυμίσω ότι είναι μια μαύρη τρύπα το, η δημοσιονομική υποστήριξη. Συμφωνώ με αυτό που είπε προηγουμένω ο συνάδελφο για ένα άλλο θέμα. Νομίζω όμως ότι οι ελπίδες που έχουν ε, εναποτεθεί στη δημοσιονομική υποστήριξη πραγματικά έχουν ε, επαληθευθεί. Καταφέραμε να κερδίσουμε το στοίχημα και μια τελευταία παρατήρηση στην οποία σχεδόν απαντήσατε. Είπατε ότι δεν υπάρχει πάντοτε κατηγορηματικό όχι σε σχέση με το αν υπάρχει κίνδυνος. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να γίνει διαχείριση κινδύνου, ευφυή μάλιστα. Γι' αυτό πιστεύω ότι στους όρους και τις προϋποθέσεις της αξιολόγησης αυτής, να έχουμε υπόψη μας τη γενική εικόνα Και κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. εγώ προτιμώ ένα σύστημα που αποκαλύπτει ένα πρόβλημα, μια δυναμία ε, για ένα σημείο, από ένα σύστημα που ποτέ δεν δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα και εσφάλματα. Υπάρχει φυσικά ένας κίνδυνος, αλλά η γενική τάση νομίζω κανένα δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι είναι αύξουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Χάουτελα, ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Μανσερβισή, και εγώ πιστεύω ότι η δημοσιονομική υποστήριξη είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο το 2012 αρχίσαμε να, το, να αποκαλούμε τις συμφωνίες συμβάσεις ε, χρηστής διακυβέρνησης, ε, τομεακές ή γενικότερες. Νομίζω ότι, όπως ε, μας είπατε, υπάρχουν πλέον ε, καλά ε, θετικά αποτελέσματα και για την εκπαίδευση και για τη δημόσια υγεία και για τη διαχείριση των ε, εθνικών πόρων, για την εξάλληψη της διαφθοράς, γιατί μας παρουσιάσατε μια σημαντική γραφική παράσταση, πολύ ενδιαφέρουσα. Δύο ερωτήσεις έχω εγώ. Ξέρω ότι στι αναπτυσσόμενε χώρε ε, υπάρχει ε, στο πλαίσιο του συντονισμού των δωρητών υπάρχουν ομάδε εργασία ε, για τη δημοσιονομική υποστήριξη. Έχετε εσεί άποψη σε σχέση με το πώ λειτουργούν, γιατί ξέρω ότι έχουν υπάρξει περιπτώσει κατά τι οποίε θυμάμαι στην Τανζανία μια φορά, ήταν απαραίτητο να γίνει αναστολή τη δημοσιονομική υποστήριξη γιατί υπάρχουν ισχυρισμοί διαφορά που έπρεπε να διερευνηθούν και νομίζω ότι υπήρχαν κάποια αποτελέσματα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι δωρητέ που συμμετέχουν στη δημοσιονομική υποστήριξη να συνεργάζονται και μερικές φορές να λένε ότι τώρα έχει γίνει παραβίαση της σύμβασης. Δεύτερη ερώτηση, κριτήρια. Ε, δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά, αλλά αν κατάλαβα καλά δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με το σε ποια ε, περίπτωση ε, ισχύει η δημοσιονομική υποστήριξη μόνο όταν υπάρχουν χρήματα ή υπάρχουν μια, υπάρχει μια σειρά κριτηρίων. Και εσείς πώς αξιολογείτε ότι μια κατάσταση είναι επαρκής για να χρήζει δημοσιονομικής υποστήριξης. Jean-Luc, ευχαριστώ πολύ για το θέμα μας αυτό της δημοσιονομικής υποστήριξης νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε δύο πράγματα. Εγώ έχω μετά από τρία χρόνια τη υποστήριξη ε, του προπολογισμού, είναι η υποστήριξη του, των οικονομικών. Δεν ε, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα εντάξει, μπορεί να είναι σε μερικέ περιπτώσει ε, αναποτελεσματική, γιατί αν ένα κράτο είναι αναποτελεσματικό για κάποιο λόγο δεν δουλεύει. Επίση, υπάρχει το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επειδή έχουμε αυτέ τι δυσκολίε. δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια χώρα χωρί να υπάρχει κράτο, πρέπει να αναπτύξουμε τα μέσα. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε ω προ την ε, δημιουργία ταμείων είναι ένα σωστό μέσο. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε το κράτος συμπεριλαμβανομένη της εφαρμογής των έργων, των ε, projects. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα ταμείο στο πλαίσιο του κράτους με ένα διπλό κλειδί, από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την άλλη το, η κυβέρνηση, έστω σε πειραματικό στάδιο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποια έργα. Γιατί ας πάρουμε το θέμα του νερού για παράδειγμα το θέμα της υγείας. Για όλα τα έργα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα μέσως, αλλά είναι σημαντικό για να υπάρχει ένα κλίμα ευνοϊκό για, την, για το περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει νερό, αν δεν υπάρχει υγεία, δεν θα έρθει κανένας επενδυτής. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν όλοι οι φορείς σε επίπεδο κράτους μαζί να συνεργαστούν με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο, δεν θα καταφέρουμε να δημιουργηθεί αποτελεσματική ανάπτυξη. Το είπαμε νομίζω ε, θα μιλήσω κυρίως για την Κεντρική Αφρική, μια ε, χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές εκλογές, από τις πιο φτωχές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολλά χρήματα ε, και γενικώ πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να υπάρξει επιτυχία. Δεν λέω ότι πρέπει η δημοσιονομική υποστήριξη να εγκαταλειφθεί εντελώς, αλλά από την άλλη θα έπρεπε ίσως η υποστήριξη προς τις ΜΚΟ να σταματήσει να υφίσταται. Θα ήθελα πάντως να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Χάουταλα, ε, ήθελα να πω ότι έχουμε ακόμη 16 λεπτά και έχουμε ε, και την, ερώτηση των την ώρα των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι σημαντική. Ε, παρακαλώ, εξασφαλίστε ότι δεν θα μιλάνε τρία λεπτά οι συνάδελφοι αντί για δύο. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε το λόγο. Δύο λεπτά. Ακόμα, ακόμα λιγότερο χρειάζομαι. Λέει η κυρία Και εγώ θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σα στο ότι σήμερα Ορισμένε χώρε αρνούνται την αντιξιακή βοήθεια και μία από τι ε, πιο χτυπητέ περιπτώσει είναι αυτό το οποίο συνέβη μεταξύ βιλγικής κυβέρνηση και Κονγκό γιατί θέλανε να γίνει ανθρωπιστική βοήθεια η ανεπτυξιακή βοήθεια, να πάει κατευθείαν στις ΜΚΟ και τότε η κυβέρνηση είπε αφήστε την ε, δημοκρατία του Κονγκό, φύγετε και κλείστε και την πρεσβεία σας. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία με τις άλλε χώρε που ε, υπάρχει τώρα. Τρέχει τώρα αυτή και πρέπει να σκεφτούμε πώ θα τη διαχειριστούμε. Thank you. You have... Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, σε σχέση με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία χρήσιμη συνεισφορά στην απόφαση που θα λάβετε εσείς σε σχέση με το πόσα ε, χρήματα θα ε, ξοδέψετε και πώς. Είδατε ότι κατά την άποψή μου προσπαθούμε να απλοποιήσουμε κάπως το περιβάλλον Όλο και περισσότερο επενδύουμε ε, με εγγυήσει. Έχουμε συνεργασία με τον ΟΗΕ κατά τον πιο στρατηγικό ε, δυνατό ε, τρόπο και συνεργαζόμαστε και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό κάνουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική σα συνεισφορά. εσεί μπορείτε να αποφασίσετε. Ε, είναι πάντως σημαντικό όλα αυτά να συνδέονται ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση στη χώρα. Μιλήσατε για τι δημόσιε προμήθειε. Εγώ το, μίλησα, το, το είπα αυτό όταν μίλησα για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αναθεώρηση. Για το θέμα Τη διαχείριση του κινδύνου στο πλαίσιο αυτό της δημοσιονομικής υποστήριξης έχουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που είναι ένα μέσο ε, για το οποίο, το, το οποίο υπάρχει σε κάθε χώρα. Ε, αν θέλετε να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Αυτό είναι ακριβώς ε, το, το εγχειρίδιο της μεθόδου μετριασμού σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Ε, πάντως το αποτέλεσμα υπάρχει επίσης. Επομένως η διαχείριση των κινδύνων είναι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνουμε και που προσπαθούμε να κάνουμε. Για το θέμα τώρα του συντονισμού των δωρητών και την ομάδα εργασίας που αναφέρατε. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, ε, ο μεγαλύτερος δωρητής στη διμερή υποστήριξη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν διάφορες ευθύνες βέβαια και διαφορετικά καθήκοντα λόγω αυτού. Ε, δεύτερον, τα προβλήματα συνήθως ε, δεν αφορούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη ενός προγράμματος και τις προϋποθέσεις για την εκταμείευση των ποσών, αλλά κυρίως το γεγονός ε, και κάποια ανησυχία εθνικής φύσεως για τη διαφθορά, ε, για την παραβίαση κάποιων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Οπότε η διαχείριση αυτού του θέματος μερικές φορές είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν καταφέρνουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και θέλουμε να παραμένουμε και υπόλογοι για το ότι κάνουμε, να μην είμαστε και να μην υπάρχει αυτόματη σύνδεση. Δηλαδή, ε, όταν ε, ε λείπουν 2 εκατομμύρια από τα 200, ας πούμε, εντάξει, αυτό έχει μια σημασία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένο με το πρόγραμμα που διαχειριζόμαστε. Τώρα, το να αναστολούμε τι πληρωμέ 200 εκατομμυρίων σε μια χώρα σημαίνει ότι επηρεάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον προπολογισμό τη χώρα δεν θέλω να, να, να ε, υποτιμήσω τη, σημασία, απλώς σας εξηγώ τι προβλήματα υπάρχουν μερικές φορές, προσπαθούμε να έχουμε ένα διάλογο, να προσπαθήσουμε να το λύσουμε έτσι, να υπάρχουν κάποια διορθωτικά μέτρα, αλλά πάση περιπτώσει έτσι έχει η κατάσταση. Τα κριτήρια για την απόφαση, εγώ πα, παρουσίασα τέσσερα στοιχεία και στο δεύτερο, το είπε η κυρία Κιέγγε, είναι προφανώς ότι εμείς βασιζόμαστε και στην πολιτική κατάσταση, στην ικανότητα του κράτους, στην αξιοπιστία του διαλόγου. Ε, ε, μερικές φορές ε, δεν είναι επαρκή για να μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε δημοσιονομική υποστήριξη ακόμη και αν υπάρχει μια ε, αξιόπιστη μακροοικονομική σταθερότητα. Υπάρχουν μερικές χώρες οι οποίες ε, θεωρούμε ότι δεν είναι πιθανό να συμβεί αυτό που δεν είναι φυκτό να καρποφορήσει γιατί υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια. Ως προς το θέμα των ταμείων Τώρα ταμεία εκτός προπολογισμού με διπλό κλειδί, τι να σας πω, δεν είναι πάντα εύκολο. Μερικές φορές υπάρχει ε, είναι, είναι δύσκολο να λέμε ότι υπάρχει ένα κλειδί από τις Εθνικές Αρχές και ένα κλειδί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ε, εκταμιευθούν τα ποσά. Τότε θα έπρεπε όμως θέλουμε η δημοσιονομική υποστήριξη να ε, χρησιμοποιείται όταν μπορούμε να πετύχουμε πραγματικά πράγματα ε, ως προς την οικοδόμηση του κράτους, όχι εκτός του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, στην Κεντρική Αφρική υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο, όμως το να πολλαπλασιάζονται τα ταμεία, νομίζω, εκτός του προπολογισμού. δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για την ε, άρνηση του Βελγίου. Κοιτάξτε, υπάρχει υπάρχουν και κάποια πολιτικά θέματα που επισέρχονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ένα ζήτημα με την πολιτική αιρεσιμότητα γενικώ. Εμείς θέλουμε να ε, παραμένουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε και να εφαρμόζουμε το άρθρο 96. Θα πρέπει να απαντήσω ούτως ή άλλως γραπτά ε, στο, στο θέμα ε, για την πληροφορική κάνουμε μια αξιολόγηση της χώρας. Για την Αιτή. Πρέπει να δούμε ε, ποιος είναι ο ε, ισολογισμός. Γιατί μερικές φορές ε, η δημοσιονομική υποστήριξη δεν συνδέεται με αυτές τις τέσσερις ε, ε, προϋποθέσεις που ανέφερα. Υπάρχει και το θέμα των αποτελεσμάτων. Υπάρχει λοιπόν μια αλληλοεπικάλυψη των δύο επιπέδων. Ε, είναι όντως συνεπής ε, στη χρήση του δημοσίου χρήματος ε, για να υπάρξει ανάπτυξη ή για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ πάντως να σας δώσω κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κατάσταση για την ώρα είναι υπό έλεγχο. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα περάσουμε αμέσως στον γύρο των ερωτήσεων. Έχουμε μια ερώτηση της Χάιντι όσον αφορά την χρηματοδότηση της υδροδότησης στην Κένια. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάουσποτ. Προφανώς ο Γενικός Διευθυντής θα μπορούσε να διαβάσει την απάντηση αλλά θα τον εκπροσωπήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων στην ε, Κένια. Και διερευνούμε τα όσα διαδραματίστηκαν την κυβέρνηση, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. Όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να σας πω ότι μία ανεξάρτητη έρευνα που έγινε από την ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το γραφείο της Amnesty International στην Κένια, ε, με τη συνδρομή των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται υπό προπαρασκευή και θα σχολιάσει σύντομα. Η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προγράμματος θα ξεκινήσει ε, εξετάζοντας ζητήματα ιδιαίτερως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απόφαση της περίπτωσης Όγκια της Αφρικανικής Επιτροπής, ε, που, απόφαση που βγήκε το Μάιο του 2017 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιωμάτα. Ε, η Επιτροπή κάλεσε την κυβέρνηση της Κένια να συμμορφωθεί ε, με το διεθνές δίκαιο που προβλέπει ότι οι αυτόχθονες έχουν το δικαίωμα στις διαχείριση της δικής τους γης και των δικών τους υδάτων. Ε, σε, μια, σε ένα δεύτερο σημείο της ερωτής, η Επιτροπή συμφωνεί με μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση σε συνεργασία με μια ομάδα ε, τοπική, ε, τοπική ομάδα συνδρομής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναστείλει τη χρηματοδότηση μέχρι να υπάρξει μία πρόοδος όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και θα προστρέξουμε στις ε, δυνατότητες διατησίας προκειμένου να βρούμε μια ειρηνική να καταλήξουμε σε μια ειρηνική διευθέτηση των ε, προβλημάτων. Heidi. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απάντησή της σε αυτή την πραγματικά σοκαριστική κατάσταση η οποία οδήγησε σε μια κατάσταση όπου η, Επιτροπή ανέστηλε το πρόγραμμα εδροδότησης. Το θέμα μου είναι το εξής. Δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε κανένα πρόγραμμα ε, περιβαλλοντικής φύσεως που αφορά την κλιματική αλλαγή εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδους ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά γνωρίζετε ότι η συζήτηση ε, εξαπλώνεται ε, όσον αφορά την μακροπρόθεσμη βοήθεια που δίνει η Φιλανδία στον τομέα της δασοκομείας στη Κένια. Και σοβαρές ανησυχίες εκφράστηκαν όσον αφορά την αξιοπιστία της ε, υπηρεσίας δασοκομείας της ε, Κένιας ε, προκειμένου να, όσον αφορά την έρευνα, τη διαρεύνηση αυτής της υπόθεσης και το κατά πόσο υπάρχει, υπήρξαν περιστατικά θανάτωσης των μελών της αυτόχθονης ε, κοινότητας. Πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της δασοκομικής ε, υπηρεσίας στην ε, Κένια ή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε τι γίνεται είτε εκεί είτε σε άλλες ε, χώρες, στην Κένια είτε αλλού. Ευχαριστώ. Είναι σωστό ότι η περίπτωση αυτή θα έπρεπε να έχει επιπτώσεις ε, ε, για όλες τις χώρες, τη Φιλανδία αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις υπηρεσίες δασοκομείας και βεβαίως ε, υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις και για τις εσωτερικές υπηρεσίες της ε, Κένιας. Γιατί τους τελευταίους μήνες είχαμε σε στενή επαφή ε, με τις υπηρεσίε αυτές και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πράγματι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο παρακολούθησης, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των εταίρων μας εκεί. Και αν ε, δεν έχουμε πλήρη ικανοποίηση ε, δηλαδή την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να εκταμιεύσουμε τα χρήματα του προγράμματος αυτού. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, υπάρχει μια δεύτερη ερώτηση που αφορά τη δημοσιονομική υποστήριξη προς την ΑΕΤ. Την είχε υποβάλει ερώτηση ο Νόρμπερτ κυρία Αντρίασεν της Επιτροπής. Reply that we have provided and uh, available. Πω, τι απαντήσαμε και αν έχετε επερώτηση, διευκρίνηση κλπ. Ό,τι θέλετε. Είπαμε ότι πρώτη για τη φτωχότερη χώρα εκεί. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη, ακόμα πλήσεται για αποθεομηνίες όπως το 16 από κάποια καταιγίδα η πολιτική είναι σε αναταραχή είχαμε το Φεβρουάριο την ε, εκλογή γενιάλψη κρατών από τον πρόεδρο Μογής To slow down a little bit. Ο πρόεδρος παρακαλούμε λίγο πιο αργά Χωρίς μικρόφωνο τώρα και υπήρχε εμπλοκή στην εκλογή του Πρόεδρου τώρα το Φεβρουάριο του 2017 ανέλαβε τα του ο νέος Πρόεδρος και έχει επίσης ένα θεματολόγιο μεταρρύθμισης και η αναπτυξιακή συνεργασία για τη χώρα ε, είναι ακόμη πάρα πολύ προβληματική και η υλοποίηση των προγραμμάτων εμποδίζεται από μια σειρά φραγμών και όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη και Ανάλογα κάνουμε και εμείς τη μεσονομική υποστήριξη με μια σειρά συμβάσεων για την ανασυγκρότηση του κράτους ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τη βασική λειτουργία του κράτους. Σαφώς έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με αυτές τις ε, συμβάσεις. Ε, Μάρτιο του 2014 με Μάρτιο του 2018 είναι σχετική διάρκεια και είπαμε ότι έχει ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογο, ο οποίος δημιουργεί το πλαίσιο για τον πάγιο μόνιμο διάλογο με τις αρχέ της χώρας κατά την διάρκεια της σύμβαση του προγράμματο και επίσης υπάρχει η οικονομική βοήθεια ούτω ώστε να υποστηριχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και έχουμε συγκεκριμένε δόσεις, μεταβλητέ, οι οποίε καταβάλλονται εάν τα τέσσερα κριτήρια τη επιλεξιμότητας πληρούνται και τα αξιολογήσαμε θετικά κατά το πρόγραμμα όπου 84 εκατομμύρια σε τέσσερις δόσεις εξετάμιευσαν και όλες αυτές οι δράσεις αφορούσαν τις επιδόσεις σε σχέση με τα κριτήρια για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών, της ε, διοίκησης και της παιδείας στη χώρα. Αυτοί η αυτά τα κριτήρια καλύφθησαν εν μέρη και είχαμε 30 εκατομμύρια και 8,6 εξ αυτών τελικά εκταμιεύθηκαν. Το πρόγραμμα επίσης προβλέπει και τεχνική αρρωγή ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις θεσμικές λειτουργίες της χώρας σε σημαντικά υπουργεία, οικονομικά, διαφθορά, παιδεία και Έχουμε κάποια παραδείγματα συγκεκριμένων ε, επιτευγμάτων, το ότι έχουμε τώρα ε, δομικό διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και αυτό αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης έχουμε τώρα πολυμερή διάλογο συντονισμού των ε, δωρητών. Όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσιονομικών και θεσπίστηκαν κάποιοι νόμοι που ορίζουν τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων. Σε διάφορα υπουργεία έχουμε συστήματα αξιολόγησης επιδόσεων και υπάρχουν διαφορά μεταξύ της διαφθοράς τα οποία υιοθετήθηκαν. Πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς του 2014 και United Λύτου σχετική μονάδα. Επομένως, συγκροτήθηκε και αυξήθηκε ε, κατά 58% το 2016 προοικοδότηση αυτή της υπηρεσίας. Και έχουμε πάνω από 60% των ε, δασκάλων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υποστηρίχθηκαν με άδειε ε, δασκαλίας 30% επίσης έγινε αύξηση των φόρων το 16 και το 17 και αρχές του 17 είχαμε 30% αύξηση του φόρου εισοδήματος επίσης για την κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο ήταν δεύτερο ήμιση της ερώτησης, ε, είχαμε τη συγκρότηση ενός εργαστηρίου το Φεβρουάριο του 2017 σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Συνένεση για τους βασικούς τομείς συνεργασίας και είχαμε επίσης ομάδες εργασίας με την κοινωνία των πολιτών και συζητήθηκε το τι έγινε με το ενδεικτικό πρόγραμμα στη χώρα από το Ταμείο Ανάπτυξης, EDF. Έτσι γίνανε επομένω οι εκταμιεύσεις ανάλογα με, τα, με τις επιδόσεις συμμετείχουν στον διάλογο όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανώσεις, η κοινωνία και δεν άλλαξε τίποτα από αυτό το ενδεικτικό πρόγραμμα μέσω της μεσοπρόθεσμης αξιολόγηση. Αυτά. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Νόρμπερτ, έχεις ζητήσει το λόγο. Ναι, από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την απάντηση της ερώτησης. Θα ήθελα να πω κάποια επιπλέον πράγματα το σκεπτικό μας. Ε, είχαμε πάει με κάποιους συναδέλφους επί τόπου και είχαμε μια διαφορετική εντύπωση όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση ιδιαίτερος. Αλλά ε, και είχαμε κάποιες εκθέσεις από ΜΚΟ που βρίσκονται εκεί και ηχούν, ακούγονται διαφορετικά από αυτά που παρουσίασε τώρα η Επιτροπή. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω την προσοχή στο εξή σημείο. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αρνείται δημοσιονομική υποστήριξη σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αυτή είναι μια ένδειξη για το που θα πρέπει να θέσουμε τα ερωτηματικά. Και όσο μιλάμε για, όταν μιλάμε για χρηστή διακυβέρνηση, βλέπουμε ότι δίνεται περισσότερο χρήματα για τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα στην ΑΕΤ από ότι για το συνολικό σύστημα υγείας στη χώρα. Νομίζω ότι αυτές είναι ερωτήσεις όπου θα αναμέναμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις από την Επιτροπή. Okay, you have a Έχετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ για την ε, επιπρόσθετη πληροφορία. Έχουμε επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην ΑΕΤ και αυτό είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς Έχουμε βεβαίω αναλύσει τον προπολογισμό του 2017 και είδαμε κάποιες ανησυχητικές τάσεις όσον αφορά την κατανομή των χρημάτων. Αναφέρατε το ζήτημα του τομέα υγείας και τις δαπάνες εκεί. Τα θέματα αυτά προσπαθούμε να τα δούμε συστηματικά στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που έχουμε από τη μία πλευρά με την κυβέρνηση και από τους άλλους ε, δωρητές από την άλλη και στο πλαίσιο αυτής της κοινή πλατφόρμας ε, προσπαθούμε να υπάρξει μια μόχλευση των σημαντικών αλλαγών στην ε, δημόσια, δημοσιονομική, στη δημοσιονομική διαχείριση Παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Νόισερ. Είχαμε πάει στην ΑΕΤ και είδαμε ότι τα πέντε δις που είχαν δοθεί για την, ε, ως βοήθεια για τον σεισμό δεν έφτασαν πολλά στους πολίτες. Μας έδειξαν κάποια προγράμματα, κάποια project τα οποία, ε, των οποίων η ουσία είναι αμφισβητήσιμη και όταν μου είπαν πόσα χρήματα μπήκαν σε αυτά τα project ε, δεν μου δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση. Πιστεύω θα πρέπει να τονίσουμε την τελευταία απάντηση της Επιτροπής. Θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι γίνεται με αυτά τα χρήματα γιατί και το ελεγκτικό συνέδριο ε, δημοσίευσε μια έκθεση που περιλαμβάνει πολύ αυστηρή ε, κριτική για την IT. Τώρα, Πρόεδρος, περνάμε στα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Ωραία, λοιπόν. Η προσεχή συνεδρίαση είναι 19η Φεβρουαρίου, 3 το μεσημέρι, μέχρι τις 6.30 και 20 Φεβρουαρίου, 9 το πρωί, μέχρι 12.30 και 2.30 το απόγευμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους διερμηνείς και πάλι για την συνεργασία τους.